είναι το θέμα μας ε, υπαριθμών 9 στην ημερησία διάταξη. Και συμφωνήσαμε για ένα σχέδιο επιστολής προς την Επιτροπή. Και η κυρία Καλβίνια, την οποία την χαιρετώ που ήρθε στην συνεδρίαση, ε, μας λέει ότι θα πρέπει να προσέξουμε πολύ τι γίνεται με τις πληρωμές. Και θέλουμε να υπάρχει κάποια αξιολόγηση, όχι μόνο όσον αφορά τον ισολογισμό των ε, ε, πληρωμών του 2013 όσον αφορά το, τον τίτλο 2 αλλά το σύνολο των τίτλων κεφαλαίων και επίσης τη σχέση μεταξύ 2007, 2013, 2014 και επίσης θα πρέπει να γίνει ένας ρεαλιστικός για μια περίοδο που δεν σταματά το 2016. Γιατί? όλα μας βεβαιώνουν ότι τα 21 δις για το 2015 και μετά όλα αυτά αναγκαστικά πρόκειται να μας οδηγήσουν σε ένα σωρό ε, απλήρωτους λογαριασμούς για πιο μετά. Η δεύτερη απόφαση αφορά κάποιες ε, ειδοποίησεις της 24ης Απριλίου 4 Μαΐου από την Επιτροπή ούτως ώστε να μπορέσουν να προσλάβουν κάποιους ειδικούς συμβούλους και ανταλλαγή απόψεων σύμφωνα με το άρθρο 123 για το καθεστώς το οποίο αφορά ε, τους ε, λοιπούς αντισυμβαλωμένους με την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόκειται για κάποιες θέσεις που εμείς ζητήσαμε και ότι ζητούμε περισσότερες πληροφορίες. Πολύ λακωνικός ο τίτλος. Θεωρήσαμε πολύ σύντομος για να μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε. Οπότε ας συνεχίσουμε τώρα τις εργασίες μας από εκεί που σταμάτησαμε το πρωί, δηλαδή να δούμε ε, τον διορθωτικό προϋπολογισμό του διορθωτικό προϋπολογισμό αριθμών 3 για το 2015 για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκαρδιθάμπολ. Όμως, λέει η κυρία Γκαρδιθάμπολ, πρώτα πρώτα παρουσιάσει η Επιτροπή το διορθωτικό προϋπολογισμό. Η κυρία Καλβίνη θα σας παρουσιάσει αυτόν τον τρίτο διορθωτικό προπολογισμό. Η κυρία Διευθύντρια έχει το λόγο. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Et so uh, I will I will turn to to English if you allow. The first. Να σας τα πω στα αγγλικά. Αυτό το σχέδιο του διορθωτικού προπολογισμού αφορά τη χρήση 2014 και όπως γνωρίζετε Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η εργασία όταν οι λογαριασμοί κλείνουν από την προηγούμενη χρήση. Ίσως είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι το γεγονός του ότι υπάρχει πλεόνασμα δεν σημαίνει ότι θα, μπορούσαμε να έχουμε δαπανίσει περισσότερα το 2014. Και οι ικανότητες κάλυψης των πληρωμών ορίζεται από τα εξής δύο πρώτα-πρώτα κατά πόσον ε, υπάρχει ρευστό σε μηνιαία βάση. Και αυτό καθορίζεται από τους ιδίους πόρους που προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Κάποιους μήνες μέσα στη χρονιά δεν αρκούν οι ίδιοι πόροι, δεν αρκετό το ρευστό και επομένως έχουμε περιορισμένη δυνατότητα πληρωμών. Συνήθως πρόκειται για τους πρώτους μήνες του έτους. Όμως, υπάρχει και κάτι άλλο που μας περιορίζει, που δεν είναι θέμα του ρευστού είναι το κατά πόσον έχουμε τις πιστώσεις πληρωμών όπως τις έχουν εγκρίνει οι αρχές του προϋπολογισμού. Το 2014 οι αρχές του προϋπολογισμού είπαν ποιο είναι το, όριο των πιστώσεων πληρωμών. Και το ότι υπήρχε παραπάνω, παραπάνω έσοδα, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν να πάνε τα θεσμικά όργανα παραπέρα από την έγκριση. Και εδώ πέρα έχουμε τα εξή δύο στοιχεία γι' αυτό το πλεόνασμα Γίνεται στις πληρωμές που για τον ΑΒ λόγο δεν θα μπορούσαν να γίνουν πριν το τέλος του έτους. Και θα πρέπει να σας αναφέρουμε ότι παρά το ότι εγκρίθηκαν αργά το Δεκέμβριο ε, τα σχέδια του προπολογισμού, ε, εκατομμύρια για πληρωμές, 4 δις δηλαδή ευρώ πληρώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Και ο προπολογισμός εκτελέστηκε σχεδόν 100%. Τώρα, όσον αφορά τις δαπάνες, ε, είμαστε πολύ χαμηλά, ίσως πιο χαμηλά από ό,τι όλα τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει όμως και άλλο ένα πιο σημαντικό στοιχείο αυτού του πλεονάσματος. Είναι το επιπλέον εισόδημα, το οποίο μπήκε στον προϋπολογισμό μετά τους τελευταίους διωτικούς προϋπολογισμούς. Είναι τόκι και πρόστιμο. Επίσης υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο το οποίο αφορά τις, τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Όσον αφορά επομένως την ισοτιμία του ευρώ, όλες αυτές οι μεταβλητές μας οδηγούν στο πλεόνασμα 1,43 δις. Ε, το, το, πλεόν ε, τα πλέον έσοδα. Και σύμφωνα με τον δημιουργικό οικονομισμό αυτά πρέπει να μπουν στον προπολογισμό φέτος ούτως ώστε όλα αυτά να ψωρευτούν, να προσθεθούν στο τμήμα του προπολογισμού που αφορά τα έσοδα. Ό,τι άλλο θέλετε να σας το ξεκαθαρίσω. Πάντως θα θέλαμε να γίνει έγκριση συντόμως χωρίς ε, τροποποίησης. Παράλληλα για τις δαπάνες έχουμε ένα άλλο, ένα άλλο σχέδιο προϋπολογισμού. Για τις θέλετε να σας τα πω τώρα. Ίσως να σας εξηγήσω με δύο λόγια. Συνεχίστε κυρία Γενική Διευθύντρια, λέει ο Πρόεδρος. Και ταυτόχρονα έχουμε τώρα το διορθωτικό προπολισμό μόνο τέσσερα το σχέδιό του. Υπάρχει μια πρόταση κινητοποίηση του Ταμείου Ελληνική. Και να δοθούν 66,5 εκατομμύρια στην Βουλγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία. Κατόπιν κάποιων θεομηνιών το 2014. Όπω θα θυμάστε, ήταν κάποιε πλημμύρε οι οποίε χτύπησαν 130.000 πρόσωπα Κάποιοι έπρεπε να εγκατέψουν τα σπίτια τους και επίσης είχαμε πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στο περιβάλλον και τις υποδομές. Οπότε με αυτή την αρρωγή θα αποκατασταθεί η κατάσταση, θα καλύψουν το κόστος διάσωσης κλπ. σε όλες τις περιοχές που χτύπησε αυτή η θεομηνία. Και εδώ θα θέλαμε να μην υπάρξουν ε, τροποποιήσεις και να εγκριθεί ταχαίως αυτό το σχέδιο ιδιωτικού προπολογισμού. Κυρία Γκάρντια Γκάρντιε Πρόεδρε ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα βέβαια να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή για τα όσα μας εξήγησε για αυτούς τους δύο διορθωτικούς προϋπολογισμούς. Όλα όσα μας είπε ήταν πάρα πολύ χρήσιμα, ιδίω για τον τρίτο διορθωτικό προϋπολογισμό, εκεί που έχουμε το πλεόνασμα, γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε. Τι είναι οι πιστώσεις ε, πληρωμών κλπ. λοιπά Τι θα πρέπει να επιστραφεί σε εισαγωγικά στα κράτη-μέλη. Όμως, δεν θέλουμε να πούμε ότι πάντα όταν υπάρχει ένα πλεόνασμα το κοινοβούλιο δεν βλέπει με καλό μάτι αυτά τα αριθμητικά στοιχεία αυτά τα ποσά που καταλήγουν στο τα πρέπει να επιστραφούν κάποια χρήματα στα κράτη-μέλη. Γιατί όπως και με άλλους προϋπολογισμούς θα πρέπει να δούμε εάν όντως θα πρέπει να επιστραφούν τα χρήματα στα κράτη-μέλη. Άρα θα πρέπει να εξετάσουμε από κοινού αυτά τα δύο σχέδια προϋπολογισμού δεν συνδέονται άμεσα και αυτόματα, αλλά απλώ γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το Συμβούλιο. Έχουμε διαφορετική ερμηνεία όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο. Στο τι πρέπει να γίνει σε αυτές τις περιπτώσεις με το Ταμείο ελληνική. Και έχουμε εδώ πέρα και αυτό το Ταμείο ελληνική θεωρεί εδώ πέρα η Επιτροπή ότι εδώ ξεπερνούμε τα περιθώρια και για τις πληρωμές και για τις υποχρεώσεις. Οπότε για το 4 θέλουμε αυτά τα 66 εκατομμύρια θα πρέπει να διατεθούν, να δεσμευτούν τέλο πάντων, ούτως ώστε να πληρωθούν στα κρατή-μέλη τα οποία θίγησαν από τις πλημμύρες. Νομίζω ότι είναι εξισορροπημένο αυτό. Τους δίνουμε κάποια χρήματα και ζητάμε αυτά τα, αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσουμε χωρίς να στρογγυλεύουμε. Ξέρουμε όμως ότι πάντοτε υπάρχει κάποια αντιπαράθεση και πέρσι επίσης στις διαπραγματεύσεις για το 2015 έπρεπε να μην αποφασίσουμε για δύο διοικητικούς προϋπολογισμούς και έτσι εκκρεμούσαν αυτοί οι δύο διότι οι του 2015. Οπότε, να εγκρίνουμε εμείς αυτούς τους προπολογισμούς, αλλά ελπίζουμε το Συμβούλιο να κάνει αυτό το οποίο πρέπει, μια που το Ταμείο Ελεγγύης είναι, είναι κάτι, είναι κάποια ποσά, ε, κάποιο ρευστό που δίνεται επιπλέον, παραπάνω και πέρα από τα ε, περιθώριο. Ευχαριστώ. Ποιος θα ήθελε να πάρει τον λόγο. Αν μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο. Α, συγγνώμη. Κύριος Μεριστάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Γιατί και εγώ είμαι συγγητής για την απόφαση κινητοποίηση ε, του Ταμείου Ελληνική για τι πλημμύρε στη Βουλγαρία, Ιταλία και Ουγγαρία. Και θα ήθελα και από τη δική μου πλευρά να δώσω πλήρη στήριξη στην προσέγγιση της ε, εισηγήτριας, κυρία Γκαρβίας Ζαντεμπάλ, γιατί νομίζω και ελπίζω ότι τα κονδύλια αυτά θα είναι καινούργια, φρέσκο χρήμα. Και για μένα είναι θέμα αρχής. Να επιμείνουμε σε θέση που έχουμε εκφράσει το παρελθόν ως κοινοβούλιο, σε πολλές περιστάσεις, ότι τα ειδικά μέσα είναι πέραν και υπεράνω των οροφών του ευρωπαϊκού προπολογισμού. Επομένω, ε, ελπίζω και περιμένω αυτή η διαδικασία να μην συνδεθεί με την ε, δημοσιονομική διαδικασία του 2016 όπως έγινε πέρσι. Ιδίω σε αυτή την ε, περίσταση, κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε καθυστερημένη υιοθέτηση της απόφασης και καθυστέρηση τη μεταβίβαση των ποσών. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ξεκάθαροι και να εμείνουμε στη θέση μας. Ότι δηλαδή πρέπει να, πάμε πέρα και πάνω από ε, τα όρια του προπολογισμού, τις οροφές. Ευχαριστώ. Κύριε Ντεγανό, ευχαριστώ. Βεβαίω και συμφωνώ με την εισηγήτρια. Όμως διερωτώ με, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να επιστρέψουμε αυτά τα χρήματα ε, στα κράτη-μέλη. Έχουμε έναν προπολογισμό, τον εκτελούμε, όχι πάντα 100% και ό,τι δεν δαπανάτε μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Διερωτώ λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την πρακτική. Εγώ θεωρώ ότι πρόκειται για ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν γίνεται να επιστρέψουν στα κρατημέλη, είναι ευρωπαϊκά τα κονδύλια. Πρέπει να μείνουν στην Ευρώπη. Ο κύριος Νοβάκοφ. Благодаря, господин Ευχαριστώ. Τα στατιστικά στοιχεία για τη Βουλγαρία είναι ξεκάθαρα. Οι ζημιές ανέρχονται σε περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ και το μεγαλύτερο μέρος ε, της ε, βοήθειας αυτής θα είναι θα αφιερωθεί για την αποκατάσταση των υποδομών και τα υπόλοιπα για την ε, παροχή μάλλον του δικτύου ίδρευσης. Όμως υπάρχει και κάτι που ξεπερνά τα αστατικά στοιχεία. 700 οικογένειες επλήγησαν σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης. Όπως είναι, είναι η πόλη της Βίζια. Φαντάζεστε τι σήμανε αυτή η καταστροφή για τους κατοίκους και ελπίζουμε αυτή η οικονομική βοήθεια να φτάσει στους κατοίκους το συντομότερο δυνατόν. Γιατί η καλύτερη βοήθεια είναι αυτή που φτάνει γρήγορα τα άτομα που τη χρειάζονται. Ελπίζουμε λοιπόν αυτός ο φάκελος ε, να προωθηθεί το συντομότερο δυνατόν. Έχοντας κατά νου την κατάσταση σε αυτές τις περιοχές. Ευχαριστώ. Ωραία, θα κλείσουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Να δώσουμε και πάλι ίσως ε, το λόγο στην κυρία Καλβίνιο. Πράγματι, ε, υπάρχει, υπήρξε μάλλον έντονη συζήτηση τα τέλη του 2014 για να πάρουμε 4,8 δις ευρώ για επιπλέον ε, πιστώσεις πληρωμών. Ουσιαστικά με αυτό το ποσό 1,35 δις έχουμε την εντύπωση ότι δεν λάβαμε 4,8 δις αλλά 3,5 γιατί στο τέλος της χρονιάς 1,35 δις τα αφήσαμε στην άκρη και επέστρεψαν ε, στα κράτη-μέλη. Είναι σαν να μας έκαναν μπλόφα ουσιαστικά. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που λέω, αλλά... Σωστό, είναι αλήθεια ότι αυτό βάζει κάποιον σε πειρασμό. Αλλά δεν δίνουμε τίποτα στα κρατημέλη τα οποία ε, δεν έπρεπε ήδη να βρίσκονται στον κόρβανά τους. Με τι να κάνουμε, έχουμε τα 25 δις ακόμα που είναι απλήρωτοι λογαριασμοί. δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες αλλά στην Ισπανία πρόκειται για κάποια χρήματα που πρέπει να μπουν στον προπολογισμό και τέλος της χρονιάς γίνεται ο ισολογισμός. Ε, αν λείπουν χρήματα πληρώνεις, αν περισσεύουν στα πληρώνουν. Γι' αυτό και κάνουμε αυτόν τον παραλογισμό. Τα κράτη-μέλη πρόκειται να ρίξουν χρήματα στον προπολογισμό, όπω ακριβώ υπολογίζεται και σύμφωνα με, υπο, με του υπολογισμού. Οπότε και αυτό ο υπολογισμό ε, πρέπει να υπολογιστεί από του ε, δασμού τελωνιακού, από τα πρόστιμα και η προσαρμογή του προπολογισμού γίνεται ακριβώ ανάλογα με το τι χρήματα δίνουν οι χώρε. Και σε αυτή την περίπτωση όμω έχουν βάλει παραπάνω πλεόνασμα. Όμως από να λέμε και εμείς ότι μια που έχουμε τα απλήρωτα θα πάνε και τα χρήματα και έτσι θα εξισορροπηθεί το θέμα. Από την άλλη μεριά βέβαια, οπωσδήποτε έχουμε τον δημοσιονομικό κανονισμό και δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τίποτα από αυτά που προβλέπει. Όμως αυτό μας εξυπηρετεί γιατί έτσι γίνεται πιο εύκολη η συμφωνία μια που υπάρχει αυτό το, ε, το, το του ενός δις Οπότε δίνουμε τα 66 από το Ταμείο Ελληνικής και αυτό βέβαια δεν πρόκειται να πειράξει την οικονομία και τους προπολογισμούς μας, οπότε θα γίνει η επιστροφή, αλλά θα πρέπει αυτό το έξτρα να πληρωθεί, αυτό το οποίο προέρχεται από το Ταμείο Ελληνικής. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι περίπλοκη συζήτηση, γιατί μας βάζει σε πειρασμό αυτή η κατάσταση. Δεν είναι θέμα cash, είναι θέμα ταμιακών ροών. Βεβαίως, δεν υπάρχει θέμα ε, καθυστέρησης, ε, όσων είχαμε, σκοπεύαμε να δαπανίσουμε για τις ε, θεομηνίες και τις φυσικές καταστροφές στη Βουλγαρία, στην Ιταλία και στη Ρουμανία, όπως ε, ανέφερε ο κ. Νορβακόφ και άλλοι. Όμω, τα 66 εκατομμύρια θα μπορούσαν βεβαίως να συνδεθούν με το 1, με τα 4,35 μάλλον. Όμως σήμερα το πρωί, κύριε Καλβίνιο, κάναμε μια συζήτηση για τη χρηματοδότηση της ε, εγγύησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. ...1,435 δις αυτό θα μας επέτρεπε να πάμε μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση χωρίς ε, να θυσιάσουμε ε, την διευκόλυνση της στην Ευρώπη ούτε τον ορίζοντα 2020. Ο κύριος Όλμπριχτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω πολωνικά. Κατά τη γνώμη μου, σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα έχουμε δύο αντίθετες προσεγγίσεις. Δύο διεφθάμενες απόψεις. Αφενός θέλουμε να ενεργήσουμε λογικά. Αυτό είναι κάτι που δύσκολα μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολιτικούς και στους πολίτες. Πρέπει να γίνονται οι πληρωμές και δεν μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή. Ή φαίνεται λογικό. Από την άλλη όμως πρέπει να ακολουθήσουμε και κάποιες διαδικασίες Έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω αν μπορεί να το ριστεί αυτό η συγκήτρια. Το θέμα αφορά τις οροφές. Ακόμα και αν έχουμε επιπλέον ε, πόρους και κονδύλια, δεν έχουμε δυνατότητα να τα αξιοποιήσουμε. Πρέπει να χρησιμοποιηθούμε με διαφορετικό τρόπο εξαιτία ε, δημοσιονομικών περιορισμών. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να διαδοθεί. Αυτές είναι οι επιπτώσεις του γεγονότος ότι είναι τόσο χαμηλά τα όρια αυτά, οι οροφές. Αυτό συμβαίνει στην πράξη. Δεν είναι μόνο ένα θεωρητικό εμπόδιο. Ως εκ τούτου η κατάσταση δεν είναι πλέον λογική. Έχουμε χρήματα που δεν μπορούμε να δαπανίσουμε επειδή οι οροφές είναι πολύ χαμηλές. Είναι, θα είναι και ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα κατά την ε, αναθεώρηση ε, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Τα κάτι μέλη θέλουν να κατεβάσουν και άλλο τα όρια αυτά και πάλι θα, θα μπαίνουμε σε αυτόν τον φαύλο κύκλο. Όσο χαμηλότερα είναι τα όρια, τόσο μικρότερα θα πανίσουμε τα κονδύλια μα. Αυτό συμβαίνει και με το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έχουμε και πάλι αυτόν τον φαύλο κύκλο. Ευχαριστώ κύριε Μαδαγκάλ. Εν συντομία. Θα ήθελα απλώς πρόεδρε να σας πω ότι συμφωνώ με την κυρία Γκαρδία Και άκουσα όλα αυτά τα ξεκάθαρα και εκπαιδευτικά που μας είπε η κυρία Γκαρδία Οπότε όλα αυτά σημαίνουν ότι το πλεόνασμα δεν προέρχεται από αδυναμία να δαπανίσουμε τους πόρους αλλά από κάποια έξτρα έσοδα. Άρα δεν πρέπει να δούμε τρόπο να, να ε, αξιοποιηθεί καλύτερα η ετήσια εισρωή κάποιων εσόδων και να δούμε μετά πώς λέω γι' αυτό αντισταθμιστικά όπως είπε η αγκαρδια Θάμπερτ. Το θέμα είναι το εξή. Αν πάντοτε η προσαρμογή γίνεται επί τη βάση των εισφορών των κρατών μελών, τότε είμαστε καταδικασμένοι στο να κάνουμε κάτι το οποίο είναι άσκοπο που συζητάμε και συζητάμε. Και έτσι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να εφαρμοστούν κάποια κριτήρια που να έρουν ε, αυτή την αντίφαση, τη, τη σύγκρουση μεταξύ των, του πλεονάσματος από την μία μεριά και την άλλη μεριά των όσων δεν έχουμε πληρώσει. Αυτά που μας εξήγησε και ο Πρόεδρος. Σε σχέση με τις στατικές επενδύσεις, με το εγγυητικό ταμείο για το σχέδιο Γιούνκερ κλπ. Και 1.800 εκατομμύρια τώρα, ένα δις δηλαδή 800 θα γυρίσουν στα κράτη-μέλη. Οπότε έτσι θα πρέπει να δούμε το πώς θα επιλύσουμε με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα. Ευχαριστώ. Δεν ζητά κανεί άλλο το λόγο. Επομένω, να δώσουμε το λόγο στην κυρία Καλίνιο. για να μας πει τη δική της ε, προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτό το πλεόνασμα και τη χρηματοδότηση του Ταμείου Αλληλεγγύης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να απαντήσω στα διάφορα θέματα προβάλλοντας τρία σημεία. Πρώτο, συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με εκείνους εξημών που τονίσατε ότι υπάρχει ανάγκη κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης, που υποτίθεται ότι είναι ένας μηχανισμός ταχείας αντίδρασης. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να κινητοποιείται, να δραστηριοποιείται σε όλο το έτος και είναι δυνατόν να μπαίνει σε ένα πακέτο με τις διαπραγματεύσεις για το σχέδιο προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, όπως έγινε και πέρσι. Συμφωνώ με την κυρία Γκάρδια Σαβάλ και άλλους ε, συναδέλφους σας ότι το Ταμείο αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο ιδιαίτερης μεταχείρισης και να είναι άνω των ε, κατοφλίων του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερους μηχανισμούς και αντίθετα με αυτούς, μιλούμε τώρα και για άλλους ε, μηχανισμούς, δεν μιλούμε για ειδικού μηχανισμούς, μιλάμε για προγράμματα εν τέλει, που έχουν περιληφθεί μέσα στα, στις οροφές του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και από όπου και να πάρουμε τα χρήματα, τα, οι οροφές πληρωμών υπάρχουν. Για όλη την περίοδο. Άρα δεν μπορούμε να επινοήσουμε διαφορετικούς πόρους από το πουθενά. Θα χρειαστεί να γίνει μετακίνηση από άλλα τμήματα του προϋπολογισμού. Τα έσοδα και το πλεόνασμα δεν έχουν σχέση και πάλι με την ικανότητά μας να τα ε, καταβάλουμε στο ΕΦΣΑ ή στο ΣΕΦ e ή στον ορίζοντα 2020. Όπως είπα και πριν, τα ανώτατα ποσά που μπορούν να δαπανηθούν ανέτος καθορίζονται από τις πιστώσεις πληρωμών και όχι απαραίτητα από τα ταμιακά διαθέσιμα που έχουμε. Και έρχομαι στο τρίτο σχόλιο για την ερώτηση του κυρίου Μαδραγάλ και όπου θεωρώ ότι είναι αλήθεια πράγματι ότι κάθε χρόνο καλούμεθα να κάνουμε προσαρμογές σχετικά με τα έσοδα. Προσπαθούμε να προβλέψουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ορισμένα πράγματα δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν στη φάση σχεδιασμού του προπολογισμού. Για φέτος έχουμε έξτρα έσοδα από τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους. Γιατί? Γιατί η ευρωπαϊκή οικονομία, βέβαια εδώ κάνω κάποιες εικασίες, έχουν περισσότερες εισαγωγές. Η αξία των εισαγωγών είναι μεγαλύτερη. Επομένω, τα έσοδα από τα τελωνία είναι υψηλότερα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Μερικές φορές υπερβαίνει τι προβλέψει μα, άλλε φορέ μένει πιο κάτω. Το δεύτερο έχει σχέση με την ε, υποτίμηση του ευρώ. Πάλι κάτι το οποίο δεν, μπορέσαμε, δεν μπορούσαμε να προβλέψουμε ένα χρόνο πριν, γιατί άλλαξε και η νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τραπέζη. Δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε. Το τρίτο στοιχείο είναι τα πρόστιμα. Σωστά είπατε ότι τα ποσά που έχουμε λάβει τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν τα ποσά που έχουμε εντάξει στον προπολογισμό. Εδώ όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Ας μην είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Πριν βάλουμε υψηλό ποσό από τα πρόστιμα στον ε, προπολογισμό, διότι αυτό θα σημαίνει, όπως είπε και η Αγκαρία Σαμπάλ, ότι τότε θα ζητήσουμε λιγότερους πόρους από τις χώρες Και αν κάνουμε λάθος, τότε θα χρειαστεί να ζητήσουμε μετά, μέσα στη διάρκεια δηλαδή του δημοσιονομικού έτους, να ζητήσουμε παραπάνω λεφτά από τις ε, χώρες μέλη. Κάτι που πολιτικά είναι πιο περίπλοκο να να το πω έτσι ας πούμε, αλλά και ε, είναι και περίπλοκο διαδικαστικά. Όταν ζητήσαμε από τις χώρες μέλη να συμβάλλουν, να συνεισφέρουν περισσότερα από ό,τι χρειάζονται, τότε επιστρέφεται, όπως είναι και σωστό. Τηρούμε λοιπόν αυτή την προσεκτική στάση σχετικά με τις προβλέψεις και την εγγραφή στον προϋπολογισμό των παραδοσιακών ιδίων πόρων ή την εγγραφή στον προϋπολογισμό άλλων εσόδων, όπως για παράδειγμα από πρόστιμα. Σας ευχαριστώ, ο Πρόεδρος. Κυρία Γκάρδια Θαμπάλ, έχετε τίποτε άλλο να προσθέσετε. Καλά λοιπόν, τότε επιβεβαιώνω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων, ότι εν πάση περιπτώσει οι τροπολογίες θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο στις 5 έκτου, ότι θα τοποθετηθούμε από αυτόν στις 23 έκτου και οι δύο διορθωτικοί προϋπολογισμοί θα μπορέσουν να φτάσουν στην ε, Ολομέλεια, σε ψηφοφορία δηλαδή, τον Ιούλιο μήνα, 7ο δηλαδή. Βεβαίω υπό την προπόθεση ότι θα έχει γίνει γνωστή η θέση του Συμβουλίου. Κυρία Καλβίνιο, λοιπόν, εσείς γνωρίζετε πώς να αντιμετωπίσετε το Συμβούλιο, ζητήστε τους να υποβάλουν την θέση τους εντός των προθεσμιών. Υπάρχει πάντως επίγον χαρακτήρα για τις χώρες που περιμένουν τις αποζημιώσεις. Ακολουθεί η κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης συνέπεια των όσων ήδη συζητήσαμε και δίνω το λόγο στον εισηγητή. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όταν συζητήσαμε τον διορθωτικό προϋπολογισμό, εξήγησα τη θέση μου και το γεγονός ότι δεν συνδέω την έκθεση αυτού του διορθωτικού προϋπολογισμού με την διαδικασία προϋπολογισμού του χρόνου που θα μας επιτρέψει να κινητοποιήσουμε από νωρίς το Ταμείο για τις ε, δικαιούχους χώρες. Θα γίνει η ανταλλαγή απόψεων στη βάση του σχεδίου εκθέσεως που δεν έχουμε ακόμη. Θα διεξαχθεί λοιπόν η ανταλλαγή απόψεων στη βάση του σχεδίου εκθέσεως την επόμενη συνεδρίασή μας στις 26 Μαΐου. Και προτείνω λοιπόν να το συζητήσουμε το θέμα τότε. Ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω να γίνονται ενστάσεις στην άποψη που εκφράσατε. Τώρα σχέδιο πληρωμών. που είναι και ένα από τα θέματα που μας απασχολούν πολύ και που μας απασχόλησαν και περί τα τέλη του 2014 και που κάπως ε, σκίασε την ε, συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2015. Καταλήξαμε στη συμφωνία εν τέλει με το Συμβούλιο με ισχυρή δέσμευση ωστόσο από πλευράς τους και από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσουν στη διάθεσή μας σχέδιο πληρωμών δηλαδή μια ρεαλιστική πρόβλεψη των, ε, της ίσπραξης και της ε, διάθεσης εσόδων και των ποσών που θα πρέπει να πληρωθούν στα τέλη του έτους. Στα συμπεράσματά μας σημειώσαμε επίσης την αρχή ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα εύλογο ανεκτό ποσό απλήρω των λογαριασμών. Αυτό δεν έγινε. Ε, προβαίνουμε σε ανταλλαγή εγγράφων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε λάβει και σχετικό σχέδιο, αλλά μας μιλούν μονάχα για την ουρά του κομίτη, δηλαδή για τα υπόλοιπα, τα πληρωτέα υπόλοιπα για την περίοδο 2007-2013. Μας είπαν ότι περί τα τέλη του 2016 δεν θα μένουν παρά 2 δισεκατομμύρια. Αυτό όμως καλύπτει, αποκρύπτει και αυτό είναι βέβαια, αυτό ισχύει μόνο για το Ταμείο συνοχή. Υπάρχουν και αλλού που δεν, ε, υπάρχουν και άλλα τα οποία δεν περιλαμβάνονται και δεν περιλαμβάνονται και τα προγράμματα τα οποία έχουν αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έστω και αν χρειάστηκε να αναβληθεί η δαπάνηση 21 δισεκατομμυρίων διότι δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν οι χώρες μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχει και αυτό ο μηχανισμό που λέει ότι όσο δεν έχει ολοκληρωθεί ένα έργο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρατεί ένα 5% και αυτό μπορεί να μεταφέρεται από χρόνο σε χρόνο όσο δεν λύγει το πρόγραμμα, το έργο δηλαδή. Αυτά έχουν ενδιαφέρον, αλλά παρόλα αυτά είμαστε Επιτροπή Προϋπολογισμών. Θέλουμε να έχουμε πίνακες ξεκάθαρους που να δείχνουν τα ποσά αυτά. Συμφωνήσαμε λοιπόν με τους συντονιστές σήμερα το πρωί ότι θα απευθύνω επιστολή στην Επίτροπο κυρία Γεωργίευα όπου θα ζητώ αυτές τις διευκρινήσεις και η κοινοποίηση αυτών των ε, στοιχείων θα υπαγορεύσει και πότε θα γίνει ο επόμενος τριμερίζης μας διάλογος περί τα τέλη Μαΐου. Αν και δεν θα είναι μάλλον μια επιχείρηση απόκρυψης ας πούμε, αυτό που θέλουμε είναι να χυθεί άπλετο φως στους απλήρωτους αυτούς λογαριασμούς ώστε να ληφθούν μέτρα για να αποφευθεί αυτή η συσσόρευση χρεών που στερεί την αξιοπιστία ενός οργανισμού όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεταφέρω λίγο, αν θέλετε, ερμηνεύω λίγο τα όσα συζητήθηκαν σήμερα το πρωί. Να αποφύγουμε εν τέλει στα τέλη του 2015 να έχουμε ξανά μπροστά μας το πρόβλημα των απλήρωτων λογαριασμών. Και τη να έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή να μπορέσουμε να συζητήσουμε ε, εν ηρεμία τον προπολογισμό του 2016, ο κ. Φερνάντες. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ούτε καν χρειάζεται αυτή η συζήτηση κανονικά, διότι οι υποχρεώσεις που έχουν αναλυφθεί πρέπει να εκπληρούνται. Τα πάκτα σουν σερβάντα όπως έλεγαν οι Ρωμαίοι. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι υποχρώσεις. Άρα ούτε καν θα έπρεπε να τα συζητούμε αυτά. Είναι προφανές. Είναι πραγματικά ντροπή για, τους θεσμικούς, ε, για τα θεσμικά μας όργανα και προκαλεί δυσπιστία απέναντι στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Εμείς θέλουμε και απαιτούμε από επιχειρήσεις και ανθρώπους να εκπλούν τις υποχρεώσεις τους εντός 60 ημερών. Πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην τα τηρεί η ίδια αυτά και μάλιστα να θέτει και σε κίνδυνο και την ολοκλήρωση έργων. Αυτά προκαλούν πολύ αρνητικές εντυπώσεις στους πολίτες. οι πολίτες θα πούν, κοιτάξτε, η Ευρώπη μας ζητά όλο και περισσότερα χρήματα και δεν πληρώνει μετά τους λογαριασμούς της. Ερχόμαστε μετά και ζητούμε πάλι διορθωτικούς προπολογισμού. Και τι λέει ο κόσμος, να κοιτάξτε πάλι μας ζητούν παραπάνω χρήματα. Ενώ αυτό που θέλουμε εμείς είναι οι οι φυστάμενες υποχρεώσεις να εκπληρωθούν, τα χρέη να ξεπληρωθούν. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα πρόληψης, ώστε ποτέ να μην ξαναφτάσουμε στην κατάσταση αυτή. Να ξεπερνάμε δηλαδή το βιώσιμο όριο των πληρωμών. Και βέβαια πρέπει να καθορίσουμε και ποιο θα είναι το ποσό αυτό, η όροφη αυτή. Βέβαια, το Συμβούλιο εγκρίνει πληρωμές και μετά ζητεί την εκτέλεσή τους. Καμιά φορά έχω την εντύπωση ότι το Συμβούλιο εγκρίνει δαπάνες ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν. Αλλά συμβαίνει και να απαιτούνται οι πληρωμές αυτές. Θεωρώ λοιπόν και πάλι ότι αυτή η συζήτηση δεν θα έπρεπε καν να γίνει. Είναι πολιτικό πρόβλημα ενώ θα έπρεπε να είναι ένα απλά τεχνικό πρόβλημα που θα είχε εύκολη λύση. Ενδιαφέρει τους πολίτες να επιληθεί. Και αυτό πρέπει να είναι από τις προτεραιότητές μας για το 2016. Ενώ οι μεγάλες προτεραιότητες πρέπει να είναι η αλληλεγγύη, πρέπει να είναι η απασχόληση, η ανάπτυξη, η διασφάλιση της ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μεγάλη στόχη. Αυτά τα πράγματα απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες και αυτά πρέπει να απασχολήσουν και εμάς δεν θα πρέπει να χάνουμε το χρόνο μας για συζητήσεις. Monsieur un document aussi vide m'interpelle. Πάμε να προβληματίζει ότι υπάρχει ένα τόσο κενό έγγραφο. Θα πρέπει και η δέσμευση να μεταφράζεται σε κάποια νούμερα. Εδώ είναι μόνο λόγια. Είναι απαράδεκτο, δεν είναι δυνατόν έτσι να συνεχίσουμε το έργο μας. Άμα συνεχίσουμε έτσι θα υπάρχει Ευρώπη σε 4-5 χρόνια. Έχουμε αυτό το σύστημα τροφοδότηση του προπολογισμού. Κάθε φορά μας οδηγεί σε μια τέτοια προβληματική. Εγώ είμαι πεπισμένο φιλοευρωπαίο και νομίζω θα πρέπει κάτι να αλλάξει αυτό το σύστημα. Κύριος Μάνκα. Ευχαριστώ. parlamentov z Francúzska, zo Španielska, ktorí súčasne sú aj starostami, primátormi vo svojich štátoch a oni nám vtedy hovorili, že roky nedostávajú zaplatené faktúry za zrealizované projekty Υπάρχει ένα... Εδώ συζητούμε συγγνώμη για το τεχνικό. πρόβλημα. Ε, Επανερχόμεθα λοιπόν μετά από το σύντομο τεχνικό πρόβλημα. Προμηνών είχαμε διεξαγάγει εδώ συνάντηση με εθνικούς βουλευτές μεταξύ αυτών και Γάλλων και Ισπανών που είναι συχνά και δήμαρχοι στις χώρες τους και μας εξήγησαν ότι ορισμένοι εξ αυτών δεν λαμβάνουν τα χρήματά τους εδώ και χρόνια. Δεν τους πληρώνουν τη λογαριασμή τους. Και μερικοί δήμαρχοι και από τη δική μου χώρα έχουν αποθαρρυνθεί πλέον. Λένε ότι δεν πρόκειται πλέον να υποβάλουν αιτήσει για χρηματοδοτήσεις από τα διαφορετικά ταμεία διότι έχουν αντιμετωπίσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Έχω ζητήσει κατ' επανάληψη να γίνουν αναλύσεις σχετικά με το ποιες είναι οι συνέπειες από τη μη πληρωμή των λογαριασμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις καλύπτονται τα κενά αυτά προσωρινά από εθνικούς προϋπολογισμούς. Σε άλλες χώρες δεν προβλέπονται ωστόσο τέτοιες λύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε καλύτερα ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των καθυστερημένων πληρωμών. Γνωρίζουν οι χώρες ότι οι δήμοι αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα σχόλια αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω των καθυστερούμενων πληρωμών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να έχουμε στα χέρια μας μια ακριβή ανάλυση του τι σημαίνουν αυτές οι καθυστερήσεις στην πράξη. Merci, Monsieur Manka. Alors, plus personne ne demandant la parole. Ευχαριστούμε. Ο πρώτος δεν ζητεί άλλο το λόγο. Ίσως η κυρία Καλβίνιο θα μπορούσε να μα ε, επιβεβαιώσει. Α, ε, ο κύριος Μαραγκάλης το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Έχω μόνο δύο ερωτήματα, ούτως ώστε να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο είπατε κύριε Αρτούη και επίση αυτέ οι δύο ερωτήσει. το τώρα που μου ήρθαν στη σκέψη βρισκόμαστε ενώπιον ανεπαρκούς ενημέρωσης. Ε, δεν είναι ούτε χρονικά ε, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 δεν ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Κατά δεύτερο λόγο έχουμε όλο αυτό το τοπίο που δεν φτάνει μέχρι το τέλος του 2016 αλλά φτάνει μέχρι το 18-19 τουλάχιστον που είναι το τέλος της εντολής. Τι είναι αυτό τώρα, ένα θαύμα. Το θαύμα του 15-16 σε σχέση με το ότι θα ανακτηθούν τα, οι απλήρωτοι λογαριασμοί σε σχέση με τα προγράμματα του ίδιας περίοδου. Επίσης τελευταίο, κάπως πιο φιλοσοφικό, ποιος χρηματοδοτεί ποιον, ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών. από οικονομική πλευρά αυτά τα στοιχεία για του απλού λογαριασμού είναι ένα χρέο. Χρέο τη Ευρωπαϊκή Ένωση προ του πολίτε. Μόνο που μια που δεν είναι τράπεζε, δεν είναι στο χρηματοοικονομικό κατεστημένο, δεν μπορούν οι Ευρωπαίοι να αξιώσουν, να απαιτήσουν αυτά που τους χρωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούν επομένως ούτε να τα αξιώσουν, ούτε να έναντι αυτών κάτι να λάβουν βραχυπρόθεσμα. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Καλβίνιο. Πες μας τη γνώμη σας σε σχέση με αυτό το οποία συζητούμε. Τι γίνεται με τις πληρωμές. Και για αυτό το έγγραφο που έχετε. που είναι το θέμα της ε, αποστολής που θα διαβιβάσουμε στην Επιτροπή. Έχω απογοητευτεί γιατί εμεί καταβάλουμε μεγάλε προσπάθειε ε, για να καταρτήσουμε αυτό το σχέδιο πληρωμών και προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε αυτό το κείμενο όλε τι πληροφορίε που είχαμε και να είμαστε απόλυτα διαφανεί αλλά και ε, να εξετάσουμε δείκτες βάσει των ε, όσων προκύπτουν από τους ε, τίτλους. Στόχος μας ήταν να δώσουμε μια δίκαιη επικόνηση της κατάστασης στα τέλη του 2014 και τις προοπτικές του 2015 και 2016. Ανταποκρινόμενη στη θητεία, την εντολή μάλλον, που είχαμε στην Συμφωνία των Δημοσιονομικών Αρχών στα τέλη της περσινής χρονιάς για την προηγούμενη πραγματική περίοδο, αλλά και για την απαλυφή αυτής της καθυστέρησης, του backlog. Βεβαίως, με τα χαράς να συμπληρώσουμε και να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες. Όμως, θα επανέλθω σε αυτό. Δεν θέλω να δημιουργήσουμε ψευδείς προσδοκίες για το όσο πρέπει να περιμένουμε σε αυτό το στάδιο. Δεύτερον, θα ήθελα να επιβεβαιώσω ότι όταν μιλούμε για πληρωμές ε, και επιστώσει εξαιτία του πολιτού χαρακτήρα του προπολογισμού της Ευρώπης και της δομής των προγραμμάτων και της δομής των πληρωμών με προχρηματοδότηση, ενδιάμεσες πληρωμές ε, και καταληκτικές πληρωμές που προκύπτει από την πολιτική συνοχή. Και ο τίτλο 1 1β είναι ο μεγάλος παράγοντας προσαρμογή του προπολογισμού σε ολόκληρο το πολετές νομικό πλαίσιο. Είναι πιο σημαντική μεταβλητή σε τη φορά της και τις πληρωμές. Ο πολιτή λοιπόν αυτός χαρακτήρας μας οδηγεί σε μια κυκλική δομή του προπολογισμού. Επομένως, για αυτή τη χρονιά και την επόμενη, εάν οι προπολογισμοί επαρκούν, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και μάλλον να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι της καθυστέρηση από την προηγούμενη πραγματική περίοδο. Τα νέα προγράμματα βρίσκονται στα πρώτα του στάδια. Δεν έχουν καν εγκριθεί όλα τα προγράμματα όλων των κρατών μελών σε όλου του τομεί. Λογικά όλα θα πρέπει να έχουν εγκριθεί φέτος και μετά θα ξεκινήσει η προχρηματοδότηση. Όμω ο βαθμό που θα έχει αυτό αντίκτυπο στι πληρωμέ στον προπολογισμό για τι ενδιάμεσε πληρωμέ θα εξαρτηθεί και από τον ρυθμό εκτέλεση από τα κράτη-μέλη. Επομένω, είναι ουσιαστικά αδύνατον αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε εάν οι πιέσει στι πληρωμέ θα έρθουν κυρίω το 2018, το 2019, το 2020. Πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η καμπύλη τα, τα τελευταία χρόνια τρέχουσα ε, ε προγραμματική περίοδου. Είναι δύσκολο λοιπόν να προβλέψουμε πέρα του 2016. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, βελτιώνουμε τι τεχνικέ μα, όμω σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον ρυθμό ε, εκτέλεση του προπολογισμού από τα κράτη-μέλη. Σε ό,τι αφορά τώρα την τι προβλέψει του ρυθμού εκτέλεση, μπορεί κανεί να είναι εξαιρετικά αισιόδοξο, εξαιρετικά απεσιόδοξο. Όμω τα στοιχεία που καθορίζουν αυτό το ρυθμό είναι και πολιτικά, άλλα είναι καθαρά επιχειρησιακά, δυνατότητες δηλαδή υλοποίηση, άλλα είναι οικονομικά. Όπως έχετε αναφέρει και εσεί, είναι σημαντικός παράγοντας και δυνατότητα σε χρηματοδότηση από τα κράτη-μέλη. Επομένω, είναι φυσιολογικό να υπάρχει μια κυκλική τέτοια ε, εξέλιξη των πληρωμών και καθώς θα υλοποιούνται τα προγράμματα θα μεγαλώνουν και οι πιέσει στον προπολογισμό τα τελευταία χρόνια του ΠΔΠ. Τρίτη παρατήρηση. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τα επόμενα βήματα. Νομίζαμε ότι το καλύτερο θα ήταν να απομονώσουμε, την ε, συζήτηση αυτής της καθυστέρησης από τις ε, διαπραγματεύσεις για το 2016. Το καλύτερο λοιπόν για να γίνει αυτό θα ήταν οι δύο δημοσιονομικέ αρχές να συμφωνήσουν επί ορισμένων αρχών. Υπάρχει μια κοινή διάγνωση τουλάχιστον. Γιατί πέρυσι το μεγαλύτερο τμήμα της χρονιάς προσπαθήσαμε να κάνουμε ακριβώ αυτό, να έχουμε μια κοινή διάγνωση των προβλημάτων. Γι' αυτό πράγματι υποβάλαμε ένα σχέδιο κοινή δήλωση, το οποίο αν συμφωνηθεί από τις δύο αρχές, τα δύο θεσμικά όργανα, βάσει των τροπολογιών που θα κατέθεταν, θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση ενό τουλάχιστον κοινού οράματο για το πρόβλημα και πώ μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, χωρί να δεσμεύεται κανένα θεσμικό όργανο για τα ακριβή ε, στοιχεία, αριθμητικά στοιχεία για το 2016 και τα επόμενα έτη. Γι' αυτό σας καλώ ε, να υποβάλλετε τα ερωτήματά σας. Θα προσπαθήσουμε να τα εξετάσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Όμως πρέπει να εξετάσουμε μία κοινή λύση, περνώντας μία, από μια τέτοια κοινή δήλωση για να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με μια πιο σταθερή βάση σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση των απλήρωτων λογαριασμών. Να επισημάνω επίση ότι στο σχέδιο πληρωμών δεν ασχοληθήκαμε μόνο με τον τίτλο 1β, την συνοχή, αλλά και τα υπόλοιπα συγκεκριμένα 1α και 4. Νομίζω ο κύριος Φερνάντες το ανέφερε και άλλοι. Ότι πολλοί έχουν πληγεί από την ε, έλλειψη αυτών των ε, πιστώσεων πληρωμών επειδή υπάρχει καθυστέρηση εκεί που δεν θα πρέπει να υπάρχει ή λόγω τόκων που έπρεπε να αποδοθούν σε άμεσους δικαιούχους εξαιτία άμεσων πληρωμών τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ αυτού. Εξετάσαμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία στο σχέδιο πληρωμών. Θα θέλαμε να κάνουμε πρόταση προπολογισμού του 2016 και 2017, το οποίο να βάζει σε σωστή τροχιά αυτού του τίτλου για να μην ανακύπτει το ζήτημα της καθυστέρησης σε άλλους τομείς. Υπάρχουν αυτά τα επιπλέον στοιχεία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας τα δώσουμε αν τα επιθυμείτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στον κύριο Όλμπριχτ, θα ήθελα να πω ότι κατά τη γνώμη μας ποτέ δεν θέλαμε να περιοριστούν οι προοπτικές για το 2015-2016. Θέλουμε να υπάρχει αυτή η διαφάνεια και η δυνατότητα πρόβλεψης και προσανατολισμού. Βεβαίως είναι πολιτέ το δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι πρέπει να συνδιαλλαγούμε με, τις, με τα κράτη-μέλη και να καταλήξουμε σε διατάξεις που θα επιτρέψουν τον προγραμματισμό των λειτουργιών μας και τι συμβαίνει ε, με τις ε, πιστώσεις πληρωμών. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες, τους, τις ευθύνες του. Ιδάλλως ε, καταλήγουμε με όλα αυτά, τα, με όλους τους λογαριασμούς, με τα προβλήματα που αυτό ενέχει. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν ε, αυτό να γίνεται πιο συγκεκριμένο με, τους, ε, με τα συμβαλόμενα μέρη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι αυτή η κατάσταση. Και οι δύο δημοσιονομικές αρχές να συμφωνήσουν. Ναι, εντάξει, αλλά... Τι συμβαίνει στην πράξη, έχουμε σωστικά έναν εκπρόσωπο τύπου από την άλλη πλευρά, ο οποίο έχει λάβει εντολή από την προηγούμενη περίοδο και είναι σαν να μιλάμε στον τοίχο. Αυτό συμβαίνει. Ζητώ συγγνώμη, κύριο Σόλμπριχτ. Ευχαριστώ. Μία παρατήρηση και μία ερώτηση. Ένα σχόλιο που είναι σημαντικό για την Επιτροπή μας και είναι σημαντικό και για το, την Επιτροπή περιφορικών υποθέσεων. Αν υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στις πληρωμές, ποιο θα περιμένει αυτά τα χρήματα πολιτικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Σε κρατή μέλη, η αρχή πληρωμή καταβάλει τα ποσά στους τελικούς δικαιούχους, γιατί, για παράδειγμα, η αρχή πληρωμή μπορεί να είναι το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν περιμένει δηλαδή το, ο δικαιούχο τα χρήματα, αλλά η κυβέρνηση. Βεβαίω αυτό εξαρτάται και από την πολιτική τη κυβέρνηση, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών περιμένει να λάβει επιστροφέ. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει του τελικού δικαιούχου, εκτό και αν η κυβέρνηση αλλάξει ε, πολιτική απέναντι στου τελικού δικαιούχου. Γιατί ξέρει ότι δεν θα τα λάβει γρήγορα τα χρήματα αυτά. Πρέπει όμω να το έχουμε κατά νου. Και είναι ενδιαφέρον να γνωρίζει η Επιτροπή μα ποιο είναι η αρχή πληρωμών Ποιο περιμένει αυτά τα χρήματα, είναι σημαντικό. Και μετά, από το 24 πάμε στα 20 φέτος 2 του χρόνου. Αλλά μία θελής ε, ερώτηση. Μιλάμε για την παλιά καθυστέρηση ή για την ενδεχόμενη καινούργια καθυστέρηση. Γιατί τα, δύο που λέμε είναι για την προηγούμενη καθυστέρηση, το παλιό backlog. Τώρα όμως τι γίνεται. 16 λέμε, 2 από το παλιό και χ από, τα, καινούργιο. <laughs> Ναι, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι, μεν κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα στα παλιά, αλλά δημιουργούμε και ενό λογαριασμού, στο οποίο ξέρουμε πώ θα πληρώσουμε. Κύριε Καρβινιό. Ευχαριστώ. Δύο σχόλια για αυτά τα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Ποιος πλήττεται. Πέρυσι, εξαιτία τη έλλειψη πληρωμών, πιστώσεων πληρωμών, προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τι ζημιέ. Ουσιαστικά δηλαδή κάναμε μια ενεργό διαχείριση πληρωμών όπω την αποκαλούμε. Η κάθε γενική διεύθυνση προσδιορίσε προτεραιότητε σε ό,τι φάση πληρωμέ. Για παράδειγμα, η ιεραρχήσαμε μας προτεραιότητα τη συνέχιση των προγραμμάτων τον περιορισμό των, ε, της ζημιάς στην πραγματική οικονομία. Δηλαδή να πληρώνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πριν από άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Τον ιδιωτικό τομέα πριν από τα κράτη-μέλη. Να πληρώνουμε τα κράτη-μέλη υπό πρόγραμμα διάσωσης πριν πληρώσουμε τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τέτοιου είδους μέτρα έχουν λάβει οι επιμέρους ε, αρχές ε, αδειοδότησης για να περιορίσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο στους τελικούς δικαιούχους. Γι' αυτό και σε ό,τι αφορά το οικονομικό κόστος για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, όπως θα δείτε στην ετήσια έκθεση, το κόστος λοιπόν είναι πολύ περιορισμένο σε ό,τι αφορά το επιτόκιο των καθυστερημένων πληρωμών, γιατί προσπαθήσαμε να περιορίσουμε τις τελικές καθυστερήσεις στους τελικούς δικαιούχους. Τώρα, κατά πόσο υπήρξε προκαταβολή από τα κράτη-μέλη στους τελικούς δικαιούχους εξαρτάται από το κράτος μέλος. Άλλοι κάνουν προκαταβολές, άλλοι όχι. Εμείς δεν έχουμε λόγο σε αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά εμά πάντω και τι άμεσε πληρωμέ, προσπαθήσαμε να αρχίσουμε προτεραιότητε, ούτω ώστε να διασφαλίσουμε κατά μέγιστο, στο μέγιστο δυνατό βαθμό ε, τη συνέχεια των προγραμμάτων και να περιορίσουμε την οικονομική ζημία. Δεύτερο σχόλιο, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, αν μιλάμε για το παρελθόν ή για την σώρευση νέου χρέους, για να το πούμε έτσι. Μιλάμε για την καθυστέρηση της περασμένης προγραμματικής περίοδου. Για την καινούργια προγραμματική περίοδο, όπως είπα, τα νέα προγράμματα θα αρχίσουν να ξεκινούν φέτος, αρχίσουν να υλοποιούνται, το 2016 θα είναι το έτος έναρξης, το 2017 λογικά θα έχουν ε, πιάσει τελική ταχύτητα, αν θέλετε. Επομένω, ε, για να σας αναφέρω κάτι το οποίο ακόμα δεν έχει εγκριθεί από ε, το Σώμα των Επιτρόπων, θα θέσουμε στο προσχέδιο του προπολογισμού τα, προγράμματα που αντιστοιχούν στα νέα προγράμματα, για να μην δημιουργείται καθυστέρηση για τα προγράμματα που ξεκινούν το 2016. Θα βάλουμε δηλαδή τι πιστώσει ε, πληρωμών για να καλύψουν τα προγράμματα που θα ξεκινήσουν το 2016. Όμως, είναι δύσκολο να προβλέψουμε πέραν του 2016. Γιατί το τι θα χρειαστούμε το 2016 θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον ρυθμό υλοποίηση των προγραμμάτων τα κράτη-μέλη. Γιατί αν καθυστερούν τα κράτη-μέλη, ο μεγάλο όγκο θα έρθει προ τα τέλη του τρέχοντο ΠΔΠ. Αυτό προσπαθούσα να εξηγήσω πριν. Αλλά βεβαίω, όταν μιλούμε για δύο δι, εννοούμε την καθυστέρηση για την προηγούμενη πραγματική περίοδο. Και ελπίζουμε ο προπολογισμό που έχει συμφωνηθεί για το 2016 είναι επαρκή για να μην δημιουργηθεί νέα καθυστέρηση για τα νέα προγράμματα. Ελπίζω να ήμουν σαφής. Το θέμα είναι πώ θα διαχειριστούμε όλα αυτά και το πώ θα καταστήσουμε του εμπλεκομένου και τα κράτη-μέλη υπόλογου, οι οποίοι θα πρέπει να δεσμευτούν σε ένα χρονοδιάγραμμα. Τι γίνεται, όλα γίνουν ταυτόχρονα. Μα δεν γίνεται τότε να καλύψουμε τις πληρωμές. Θα πρέπει ομένω τα κράτη να λάβουν τι ευθύνε του που δεν τι έχουν λάβει μέχρι σήμερα. Κύριο Μάνκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Α υποθέσουμε ότι μια χώρα πληρώνει τους δημάρχους και ταυτόχρονα δεν πληρώνει συνεισφορά στον κοινοτικό προϋπολογισμό τελικά πρόκειται για ένα κύκλο. Νομίζω χρειάζεται μια καλύτερη ανάλυση, δηλαδή ποιο οφείλει σε ποιον και ποιε είναι οι συνέπειε αυτών των χρεών. Είναι ενδιαφέρον αυτό το έργο. Δεν ξέρω τι γίνεται σε κάθε κράτο μέλο, αλλά εγώ βλέπω τι ισχύει στη Γαλλία που έχω απευθυνθεί σε όλους τους πρόεδρους ε, των διοικητικών περιφερειών για τις πληρωμές. Και μόνο μία περιφέρεια μου απάντησε σχετικά με ακρίβεια. Οι άλλες θεώρησαν ότι απλώς αποφεύγουν να λάβουν τις ευθύνε τους και μου είπε ότι προχρηματοδοτεί. Άρα θα πρέπει να γίνουν κάποιοι έλεγχοι με τα εθνικά κοινοβούλια για να δούμε ακριβώς τι γίνεται με αυτούς τους πόρους και να είμαστε σίγουροι ότι με την προσοχή και ευστηρότητα που πρέπει ελέγχουμε. Και έτσι λοιπόν θα έρθει πιο κοντά ο πολίτης στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και εγώ. Δεν είναι καινούργια αυτά. Ήσασταν πρόεδρος ε, για τις περιφέρειες. Ναι, ακριβώς πριν από δέκα χρόνια και ακριβώς προσέγγουσαν σε αυτές τις δυσκολίες. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια φτάνανε με αρκετή καθυστέρηση. Οπότε αποφασίσαμε να γίνεται προχρηματοδότηση. Προκαταβολή για όλα τα έργα που αφορούσαν την Ευρώπη. Όμως δεν είναι η δουλειά της περιφέρειας να κάνει την τράπεζα βέβαια την άλλη μεριά είναι προς το συμφέρον της περιφέρειας και του πολίτη τα έργα να εκτελούνται. Υπάρχει μια ολόκληρη τεχνική βέβαια, ούτω ώστε να αποφεύγει κανείς αυτές τις καθυστερήσεις. Γιατί σε κάθε θητεία πάντοτε υπάρχει ένα ε, διάλειμμα ούτως υπήν Ενό έτου που δεν γίνεται τίποτα. Μου συνέβη αυτό. Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα προηγούμενα έργα και δεν μπορεί κανεί να στήσει, να χρηματοδοτήσει τα επόμενα. πρόεδρο. Αυτά όσον αφορά το σχέδιο των πληρωμών. Κάτι άλλο κυρία Καλβίνια. Να δούμε μόνο ποιο ποσό είναι λογικό που να καλύπτει τους απλήρωτους λογαριασμούς. Νομίζω θα είναι πολύ συναρπαστική η επόμενη συνάντηση. Οπότε, αλεπτρώσαμε με αυτό και προχωρούμε. Κύριος Νίκ Τζάνετ, καλώς από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι επικεφαλής του Τμήματος ε, Ειδικών ε, Συναλλαγών και επίσης ο κύριος Μπόρχαρτ Σμιτ από τη Γενική Διεύθυνση ΕΚΦΙΝ. Όπως ξέρετε υπάρχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα ούτω ώστε να υπάρξει η έκδοση των ομολόγων έργων. Χρηματοδότηση από τον προπολογισμό μέχρι 31 του 2014 έγινε αυτή η δραστηριότητα και ευχαριστώ πολύ τους ε, προσκεκλημένους μας που ήρθαν για να μας πούνε για αυτό το εγχείρημα, να μας πούνε τι έγινε. Πότε δώσω το λόγο στον κύριο Νίκ Τζάνετ. Ε, we have ε, ε, come to you today with the with our presentation and Έχουμε αυτή την παρουσίαση να σας πω το πρώτο τμήμα αυτής και ο συνάδελφος Νίκ Τζάνετ από την Τράπεζα Επενδύσεων. Εγώ θα σας πω τα της Κομισιόν. Σήμερα για να σας πούμε αυτήν την εξαμηνιαία έκθεση όσον αφορά την πρωτοβουλία για τα ομόλογα έργο. Και σας ενημερώσω και σε σχέση με το ιστορικό πλαίσιο. Στη δεύτερη διαφάνεια τώρα που βλέπετε στην οθόνη έχουμε συνοψίσει την διάρθρωση, τη δομή αυτής της πρωτοβουλίας. Σας θυμίζω ότι θέλαμε να καλύψουμε τα κενά της χρηματοδότησης για τις υποδομές με επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα. Ήταν ένα πείραμα να δούμε αν αποδίδει. Πώς έγινε. Ο σκοπός είναι να παρέμβει η Τράπεζα Επενδύσεων. Να καλύψει τους κινδύνους για την χρέωση στην οποία πάει το έργο. Οπότε αυτό το μαξιλαράκι της Τράπεζας Επενδύσεων θα οδηγούσε σε μια μόχλευση με τα ε, κοινωνικά χρήματα. Παρεμβαίνει λοιπόν η Τράπεζα Επενδύσεων με την φήμη της την εμπιστοσύνη της και έτσι τα ομόλογα έργο πιο εύκολα θα μπορούσαν να πιάσουν τόπο. Βλέπετε εδώ πέρα ε, τους τομείς που καλύπτουν αυτά τα ομόλογα, ε, τα, τα διευρωπαϊκά δίκτυα, μεταφορές ενέργεια, οριζονικά, 230 ε, εκατομμύρια καταρχήν Οπότε έχουμε πολλά χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία επιστρατεύει η Τράπεζα Επενδύσεων για να έχουμε αυτού του είδους την πίστοση. Και έτσι αναδεικνύονται τα όσα μπορούν να χρηματοδοτήσουν οι ιδιώτες. Μετά έχουμε την έγκριση κάποιων ε, σχεδίων, τον τέλος του 2014 και κάποια άλλα τα οποία πρόκειται να ε, υπογραφούν φέτος και του χρόνου, γιατί όπως ε, φαντάζεστε πρόκειται για δύσκολο έργο σαν την τεκμηρίωση αυτών των ε, σχεδίων και έργων. Τώρα, έχουμε έκθεση εγγράφους. Σύμφωνα το άρθρο 140 του Δημοσιονομικού Οργανισμού προβλέπεται μια τέτοια έκθεση ε, κάθε χρόνο. Έχουμε και μια διάμεση έκθεση του 2013 και επίσης μια εξωτερική αξιολόγηση αυτής της ε, πρωτοβουλίας που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2014. Όποιος θέλει μπορεί να την ε, συμβουλευτεί και τώρα επίσης θα αναθέσουμε την σύνταξη μιας αξιολόγησης για το 2015. Η τελική αξιολόγηση για την πρωτοβουλία των ομολογών έργων. Και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε την εξέλιξη αυτών στα πλαίσια του Βλέπουμε τώρα ότι από τότε που μπορουμε να φτασουμε την εξελιξη αυτων της πλαισια του αυτή η ιστορία έχει αλλάξει το πλαίσιο πολιτικής. Αυτό βεβαίω και το γνωρίζετε γιατί η Επιτροπή σας είναι μία από τις δύο ε, κυρίως αρμόδιες ε, ή συναρμόδιες επιτροπές που ασχολούνται με το σχέδιο Juncker. Προτεραιότητά σας είναι οι επενδύσεις. Για το σχέδιο στρατηγικών επενδύσεων και για το project portal, δηλαδή την πύλη αυτήν, αλλά έχουμε επίσης και την Ένωση της Κεφαλαίου Αγοράς, το σχετικό κανονισμό και αναλύεται τώρα το τι γίνεται με την υποδομή σε σχέση με τη συμφωνία ε, της αξιοπιστίας υπαριθμών 2 θα ολοκληρωθεί αυτή η αξιολόγηση τον Ιούνιο φέτος και όλες αυτές τις προσπάθειες πανευρωπαϊκά οδηγούν στο να προσέξουμε να δούμε ποιο είναι το συνολικό επίπεδο των επενδύσεων παγκόσμια στο πλαίσιο του G20 και του ΟΣΑ όπου και εκεί ασχολούνται με το πώς θα θεωρηθεί στοιχείο ενεργητικού ε, η υποδομή με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συλλογή δεδομένων σε κάποιο είδους ε, έργα μακρόπνο και έτσι να είναι πιο προσβάσιμα όλα αυτά σε θεσμικούς επενδυτές και να μην ε, βοηθά μόνο ο δημόσιος κορβανάς αλλά να ενισχύουν και ε, οι ιδιώτες. Τώρα, να δούμε τώρα τις εξελίξεις στην αγορά. Πέρυσι σημειώθηκε ρεκόρ όσον τη δραστηριότητα χρηματοδότησης ε, των έργων. Παγκοσμίω. Ταυτόχρονα πάντως, παρά το ότι υπήρξε περισσότερη προθυμία από τις τράπεζες για μακρόπνοιο δανεισμό, παρόλα αυτά Δεν υπήρχε αρκετή δραστηριότητα από συμφωνίες και σε ορισμένους κλάδους και σε ορισμένες χώρες. Εκεί θα στοχεύσει στο να βοηθήσει το σχέδιο Γιούνκερ και από πλευρά και ζήτησης. Εδώ τελείωσα τη δική μου παρουσίαση, αλλά θέλω να σας δείξω και αυτή τη διαφάνεια. Εδώ βλέπετε τι έγινε όσον αφορά τα δάνεια αλλά και τα ομόλογα. Βλέπουμε το 2012 ανέβηκε το επίπεδο έκδοσης των ομολόγων. Σημαντική αύξηση. Και δείτε κάτω την κόκκινη γραμμή βλέπουμε επίσης ότι το 2012 είχαμε αύξηση. Οπότε η ζήτηση για ομόλογα έργου αλλά και η έκδοση αυτών εγνώρισε μια σημαντική αύξηση. Και αυτό λόγω της εν λόγω πρωτοβουλίας που προσέδωσε αξιοπιστία σε αυτό το μέσο χρηματοδότησης. Και τώρα η σκητάλη στο συνάδελφο από την ΕΤΕ. Ευχαριστώ Μπορκχαρτ. Μεγάλη χαρά μου σήμερα που μπορώ να είμαι κοντά σας για να σας πω τι έγινε με την πρωτοβουλία των ομολόγων έργου πολύ πιο ευχάριστο να μιλώ για τα όσα έχουν γίνει παρά ε, στα αρχικά στάδια που έλεγα τι επρόκειτο να κάνουμε. Έχουμε λοιπόν συγκεκριμένα επιτεύγματα και σας τα αναφέρω. Πρώτα λοιπόν και σε ό,τι αφορά τον αριθμό συναλλαγών που έχουν ήδη κλείσει, τέσσερις έχουν κλείσει μέχρι τώρα στη διάρκεια της πιλωτικής φάσης. Πρώτο στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα έργο μεταφορών ενέργειας από ε, ανεμογεννήτριες που είναι μακριά από την ακτή. Επίσης το πρώτο Greenfield Project είναι ο επίσης αυτοκινητόδρομος ε, μη 11 στο Βέλγιο. Τρίτο, υποδομής ευρέως φάσματος στη Γαλλία. Και τέλος, ανάμεσα σε αυτή την ομάδα ε, συναλλαγών είναι και ο αυτοκινητόδρομος μη 7 στην Γερμανία. Πολύ σημαντικό έργο γιατί δείχνει ποια είναι η αξία του μηχανισμού αυτού σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τις χώρες που έχουν χαμηλότερη βαθμολόγηση με αυτές που έχουν την υψηλότερη. Εκτός αυτού η τεχνολογική, μάλλον η η ε, χρηματοοικονομική τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για δύο ε, που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τον απλό λόγο ότι τα ποσά που ήταν διαθέσιμα για έργα ενέργειας είχαν εξαντληθεί ήδη από το πρώτο έργο. Δύο λοιπόν το ε, έργο αποθήκευσης αερίου Κάστορ που όπως γνωρίζετε έχει περιέλθει ξανά στην κυριότητα του δημοσίου μετά από κάποια πολύ σημαντικά γεγονότα, ε, σεισμικά γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ε, ε, ανάληψή του από το δημόσιο και άλλο έργο που συνδέει πάλι φάρμα ανεμογεννητριών ε, στην θάλασσα δηλαδή με το δίκτυο του Ενωμένου Βασιλείου. Αυτά τα αυτοί οι μηχανισμοί έχουν οδηγήσει σε 4,4 δισεκατομμύρια ε, ε, επενδύσεις από ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι, ναι. Ο, ο αναφέρεται σε πολλούς αριθμούς που τους βλέπετε στην ε, διαφάνεια. Έχουμε επίσης τώρα και για το 2015 και για 2016, όπως είπε και ο συνάδελφός μου Σμιτ, έχουμε μέχρι τέλους του 2016 περιθώριο για να κρίσουμε έργα τα οποία έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τραπεζής Επενδύσεων μέχρι πέρσι. Και αυτός αυτή η πλέον, αυτός ο αγωγός φαίνεται να είναι ισχυρός. Ελπίζω λοιπόν ότι την επόμενη φορά που θα μας προσκαλέσετε, αν μας προσκαλέσετε για να σας μιλήσουμε για την πρωτοβουλία, θα έχουμε περισσότερα έγχρωμα τμήματα στον ε, χάρτη που βλέπετε και πιστεύουμε ότι μέσα στο κύκλο ζωής του πιλωτικού ε, προγράμματος θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε έργα και στην Ιταλία, στην Ολλανδία και ε, αλλού και ελπίζω θα φτάσουμε και στην Ισπανία και στην Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα όσα έχουμε επιτύχει ως τώρα. Τρία βασικά επιτεύγματα. Και πρώτο, η πρωτοβουλία ομολόγων έργου έχει συμβάλει χωρίς καμιά συζήτηση στην επανεμφάνιση χρηματοδότησης από τις αγορές κεφαλαίου για μακρόχρονες επενδυτικές δραστηριότητε στην Ευρώπη. Το έδειξε αυτό και στη διαφάνειά του ο κ. Σμιτ. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η PBI, η πρωτοβουλία δηλαδή, έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Δεύτερο, τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία, η δηλαδή χρηματοπιστωτική τεχνολογία στην οποία βασίζεται η πρωτοβουλία έχει δείξει την αποτελεσματικότητά της για την επίτευξη των επιπέδων ε, ανύψωση των ποσών που μπορούν να συλλεχθούν από τις ιδιωτικές επενδύσεις και τρίτο και πιο σημαντικό πηγαίνουμε πολύ καλά για να επιτύχουμε τους στόχους της πιλωτικής φάσης που, προβλε... πρόβλεπε να κλείσουν μέχρι το τέλος του 2016 5 έως 7 συναλλαγές, transactions. Και πηγαίνουμε πολύ καλά όπως είπα. Επόμενη διαφάνεια τώρα. Τι γίνεται τώρα, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Δύο εξελίξεις νομίζω μπορούμε να προβλέψουμε και πρώτη. Όταν θα ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της πρωτοβουλίας στα πλαίσια της ε, διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη, θα υπάρξει και ανάπτυξη στους τρεις τομείς που καλύπτει η ε, διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί η χρηματοπιστωτική τεχνολογία και το σχέδιο Juncker επενδυτικών πρωτοβουλίων για την Ευρώπη που καλύπτει βέβαια ευρύτερο φάσμα τομέων από αυτό που καλύπτεται στην πιλωτική μονοφάση. Τέλος λοιπόν, συνοψίζοντας περισσότερο, έως τώρα έχουμε διδαχθεί τα εξής. Ο μηχανισμός όπου εφαρμόστηκε προσέφερε σημαντικά χρηματοπιστωτικά πλεονεκτήματα στις δημόσιες αρχές και έχει συμβάλει με πολύ ε, χρήσιμο τρόπο στην καθίδρυση εναλλακτικών μορφών μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Εναλλακτικών στις τράπεζες δηλαδή. Δεύτερο, ένα από τα κύρια μηνύματα που ακούσαμε ξανά και ξανά από την κοινότητα των επενδυτών είναι ότι στην ουσία τους έχει ανοίξει όρεξη για επενδύσεις σε έργα υποδομών. Και ξανά και ξανά έχουμε δει επενδυτές να ζητούν περισσότερη προβλεψιμότητα των ε, χρηματοπιστωτικών, των επενδυτικών ε, οδών και αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι και ένα από τα συμπεράσματα που θα ε, έχουμε. Και τέλος, να τελειώσω λέγοντας ότι ανεξάρτητα από τη σημασία του οι αρχές του δημόσιου τομέα εξακολουθούν να σχεδιάζουν τις δημόσιες προμήθειες εις τρόπον ώστε να διευκολύνουν πρόσβαση στα έργα αυτά από την ιδιωτική επένδυση, από την ιδιωτική χρηματοδότηση. Σαφές μήνυμα το οποίο συμβαδίζει με την ανάλυση στην οποία βασίζεται και το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Να αρκεστώ σε αυτά κύριε Πρόεδρε και βέβαια ευχαρίστως να ακούσουμε τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Μπορείτε μόνο να μας θυμίσετε τι ακριβώς έχουν όλα αυτά για τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό και πώς συνδέεται αυτό με τις γενικές διατάξεις Κάπου διάβασα 230 εκατομμύρια. 230 εκατομμύρια είναι η συνεισφορά. Αλλά ως δάνειο ή ως επιδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, τα, τα, κονδύλια του προπολογισμού που είναι διαθέσιμα είναι πράγματι 230 δις. Πρόκειται για κονδύλια από την προηγούμενη πραγματική περίοδο που είχαν τεθεί στην άκρη ε, για να λειτουργήσουν συμπληρωματικά σε τρεις διαφορετικούς φακέλους. Για ενεργειακά προγράμματα, 10 εκατομμύρια έχουμε εκεί, ένα φάκελο για τις ευρυζωνικές τηλεπικοινωνίες, 20 εκατομμύρια εκεί, και ε, μεταφορές 200 εκατομμύρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα κονδύλια αυτά λειτουργούν συμπληρωματικά ε, για τον ε, φάκελο αυτό και για τις συναλλαγές ε, στις οποίες επιστρέφεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα επιμεριστούν τώρα τα κονδύλια αυτά μεταξύ της Τράπεζας και της Ένωσης, ανάλογα και με τους κινδύνους που αναλαμβάνονται ο προπολογισμό παίρνει την πρώτη ζημιά, η Τράπεζα Επενδύσεων εναπομείνα σε ζημίε. Εμείς ελπίζουμε στο τέλος της πραγματικής περίοδου τα κονδύλια να επιστρέφονται. Όμως αυτό εξαρτάται και από το κατά πόσο υπήρξαν ζημίες υπό αυτόν τον φάκελο ή όχι. Ευχαριστώ. Ε, στον πίνακα που μας δώσατε στη σελίδα 8 έχετε δύο στοιχεία. Φαντάζομαι ότι ήταν το τμήμα των εγγύησεων. Και μετά αναφέρεται 46 στο Off the Greater Gabbard UK. Εκεί πέρα λέτε 46 εκατομμύρια και 305 είναι ε, το γενικό ποσό, το συνολικό ποσό του δανείου. Ναι, έχετε δίκιο. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον Greater Gabbard. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει ε, δώσει πιστοτικό έγγραφο ε, στο ύψος των 46 εκατομμυρίων. Δεν έχει χρηματοδοτηθεί, είναι μερική εγγύηση τώρα αυτό. Εάν είναι απαραίτητο, τότε μπορεί να αξιοποιήσει αυτή η επιχείρηση, αυτή την εγγυητική επιστολή, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει τυχόν δυσμενείς ε, συνθήκες. Μέχρι τώρα δεν έχει συμβεί αυτό. Τα 305 εκατομμύρια αφορούν την αξία των ομολόγων που εκδόθηκαν από την επιχείρηση στην αγορά και τα έσοδα αυτής της έκδοσης λειτουργούν ε, για την συμπλήρωση του χρέους. Η συνολική δηλαδή χρηματοδότηση είναι η ίδια κεφάλαια που δεν έχω σημειώσει εδώ, συν ε, το επιπλέον κεφαλαιοποίηση μέσω των ε, ομολόγων των 305 εκατομμυρίων. Και αυτό συνοδεύεται και από μια εγγυητική επιστολή από την τράπεζα που θα μπορούσε να επικληθεί η επιχείρηση εάν αυτό είναι απαραίτητο. Αυτή η συναλλαγή ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα γιατί ήταν πολύ ελκυστική η κοστολόγηση της έκδοσης ομολόγων. Ξεπεράστηκε κατά τρεις φορές λοιπόν το αρχικό ποσό που δείχνει και τον, ε, το ενδιαφέρον των επενδυτών σε αυτές τις υποδομές, τον κλάδο των υποδομών. Και η τιμολόγηση των ομολόγων ήταν τέτοια, ούτως ώστε το κύριο χρέος ήταν με τους καλύτερους δυνατούς ε, όρους. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση. Η εγγυητική αυτή επιστολή, καθώς και η έκδοση ομολόγων γίνεται σε τερλίνες? γιατί αν αυξηθεί η τιμή του της ε, λίρας της Βετανικής, τότε αυτό θα σημάνει ζημία στην αλλαγματική. Πράγματι, η εγκυτική επιστολή δίνεται σε λίρες Αγγλίας. Και αν ε, γίνει εξοποίηση της εγκυτικής επιστολής, ε, τότε το ποσό αυτό θα αντληθεί από το και σε ευρωφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η αξία του φακέλου βεβαίως και βασίζεται στην ε, συναλλαγματική ισοτιμία. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ε, τα στοιχεία, αλλά μπορούμε να σας τα δώσουμε αν σας ενδιαφέρει. Ευχαριστώ. Κύριος Κολμέλνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ομολογώ ότι η ενημέρωση αυτή, για την οποία ευχαριστώ, με οδήγησε μεγαλύτερη σύγχυση. Μιλούμε για ομόλογα έργου και διερωτώμε πρώτα-πρώτα υπό τον τίτλο «Διαφάνεια του προϋπολογισμού μας» Πού θα πρέπει να κατατάξω αυτά, δηλαδή σε μια προσπάθεια διαφάνεια του προπολογισμού. πού θα πρέπει να κατατάξω αυτά τα ομόλογα έργου. Ομολογώ ότι δεν κατανοώ καν γιατί συζητούμε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τέτοιου είδου χρηματοδοτικά μοντέλα. Βλέπω στη σελίδα 8 ότι υπάρχει ένα έργο, ο αυτοκινητόδρομο υπαριθμών 9 στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, που προβλέπεται ω έργο που θα χρηματοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό. Και διαβάζω ταυτόχρονα ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και για μια περίοδο έως 7 χρόνια πληρώνει αρνητικούς τόκους για την δανειοδότησή του. Πού βρίσκεται λοιπόν το πλεονέκτημα του χρηματοδοτικού μηχανισμού μέσου ομολόγων έργου. Μου φαίνεται ότι πάμε να μπούμε μέσα σε ένα πάρα πολύ περίπλοκο μηχανισμό που ίσως κατανοούν κάποιοι εμπειρογνώμονες, σίγουρα όχι ο απλός πολίτης. Πού κρύβεται το πραγματικό πλεονέκτημα. Γιατί δεν επιλέγονται ξεκάθαρες δανειοδοτικές δυνατότητες, ας πούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει ότι θέλει να χρηματοδοτήσει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στη Γερμανία, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ως Γερμανός πολίτης. Διαρωτώ με όμως αν είναι σωστό άψη επικουρικότητας ως Ευρωβουλευτής. Και διαρωτώ με επίσης χρειάζονται πραγματικά αυτά τα προϊόντα, διότι κάπου χάνουμε πλέον και την εποπτεία για το ποιο αναλαμβάνει ποιο κόστος και τελικώς ποιο είναι το Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σουσανή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τους ε, προσκεκλημένους μας για την παρουσίασή τους. Εγώ δεν είμαι και τόσο ενθουσιώδης με βάση αυτά τα αποτελέσματα των βιβλιοτικών προγραμμάτων. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για αποτυχία και θα σας εξηγήσω πού βασίζω αυτή την άποψη. σου μπορείτε και εσείς να μου δώσετε κάποιες απαντήσεις. Πρώτον, σε... αν είχαμε επαρκή ρευστότητα, ιδίως στις κεφαλαιογορές, και με δεδομένο το χαμηλό φορολογικό συντελεστή, πολύ πιθανό αυτά τα πράγματα να είχαν χρηματοδοτηθεί χωρίς ε, ε, την αναγκαιότητα να υπάρξουν δημόσιε εγγυησει. Επομένω, με αυτέ τι εγγύησει, το μόνο που καταφέραμε ήταν να μεταβιβάσουμε τον κίνδυνο από τον ιδιωτικό επενδυτή στο δημόσιο τομέα και στους πολίτες, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και μάλιστα σε μια χρονική στιγμή που δεν χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Εάν είχαμε επαρκή ρευστότητα, χαμηλού φόρους, με ευκολία θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθεί όλα αυτά, χωρίς τέτοια δημόσια εγγύηση. Σήμερα μιλούμε για το έργο Juncker, το πρόγραμμα Juncker, το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και επικεντρωνόμαστε εδώ στην προσθετότητα. Εδώ εγώ δεν βλέπω ακριβώς αυτό το στοιχείο, την ε, επιπρόσθετη αξία. Κάτι άλλο που ήθελα να δείξω. Τι γίνεται ακριβώς ε, κατά την χρηματοδότηση των προγραμμάτων. Κάποιες φορές είναι αμφιλεγόμενη επιλογή του προγράμματος ή επιλέγεται η αναχρηματοδότηση ενός υφιστάμενου χρέους. Δεν υπάρχει προσταθεμένη αξία σε αυτή την περίπτωση, απλώς αναχρηματοδοτούμε υφιστάμενο χρέο από παλιέ υποδομέ. Και αυτό σε καμία περίπτωση δεν είναι ο στόχο μας. Δεν δημιουργούμε έτσι κίνητρα για νέες επενδύσεις. Αυτό γίνεται με την, ε, με την δημιουργία και υλοποίηση νέων προγραμμάτων υποδομών, όχι παλιών. Το πρόγραμμα Κάστορ, όπως ξέρετε, Ε, σε μεγάλο βαθμό συνέβαλε στην αποτυχία του προγράμματος. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Έτσι πώς γίνεται η αξιολόγηση των αιτήσεων στην πρωτοβουλία αυτή. Στο Κάστρο ήταν αρκετά σαφές ότι τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε. Θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς τι ακριβώς πήγε στραβά λοιπόν. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες θα ήθελα για το εξή θέμα. Πέραν τη εγγύηση που δίνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, τι ακριβώ έχει επενδύσει η Τράπεζα Επενδύσεων σε αυτά τα προγράμματα. Γιατί πέραν των εγγύησεων έχουν επενδύσει κιόλα. Έχει επενδύσει η Τράπεζα Επενδύσεων στα ομόλογα αυτά. Περίπου 300 εκατομμύρια νομίζω. Καλό θα ήταν λοιπόν να έχουμε αυτές τις πληροφορίες ε, για να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Και τώρα που μιλώ για διαφάνεια, αυτές οι πρωτοβουλίες προγραμμάτων, και εδώ συμφωνώ με τον προλαλήσαντα, ξέρω ότι είναι ιδιαίτερα πρόκειται για περίπλοκα μέσα και εργαλεία, όλα αυτά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα, ιδίω για τον ε, μέσο άνθρωπο, δύσκολο να τα κατανοήσει κανείς. Όμως για τη διαφάνεια, τι ακριβώς ε, σκοπεύετε να κάνετε βάσει τη νέα πολιτική διαφάνεια της ERB. ίσως τα πράγματα να χειροτερεύσουν και όχι να βελτιωθούν. Και το τέλος, ο κ. Καναπιέτο, πρώην αντιπρόεδρος, είχε πει ότι θα θέλαμε να εκδώσουμε αυτά τα ομόλογα έργων για να θυματοδοτήσουμε χρέη για τη φετινή χρονιά. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε κάτι για την έκθεση για την δραστηριότητα της ε, Τράπεζας Επενδύσεων που υπεψηφίσαμε την περισμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Τι προτίθεται να κάνει λοιπόν η Τράπεζα Επενδύσεων. Θα ακούσετε τη φωνή του Κοινοβουλίου. Θα λάβετε υπόψη το γεγονό ότι δεν θέλει το Κοινοβούλιο να χρηματοδοτήσει αυτό το πρόγραμμα, αυτό το έργο. Ευχαριστώ κύριο Δενανό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Μιλήσαμε επιμακρών για τα ομόλογα έργου, αλλά δεν είχαμε συγκεκριμένη ιδέα περί τίνος πρόκειται. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το σχέδιο Juncker ε, κυρίως αφορά επενδύσεις και εγγυήσεις επενδύσεων. Επιστρέφουμε λοιπόν στην ίδια προβληματική. Να σας πω ότι κάποια προγράμματα αφορούσαν και την περιφέρειά μου και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι επέτρεψε αυτό να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα που θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί αν δεν υπήρχε αυτή η διάταξη. Ουσιαστικά μιλάμε για ε, τεχνολογίες υψηλής ταχύτητας, πολύ υψηλής ταχύτητας, ακόμα και σε γεωργικές περιοχές. Γιατί στη Γαλλία, όπως ξέρετε, είχαμε κάποιες συγκεκριμένες ζώνες που αφορούσαν μόνο τους πολύ παραδοσιακούς παρόχους και εκείνοι πήγαιναν μόνο εκεί πέρα που είχε κέρδος. Τα υπόλοιπα, την ύπεθρα την είχαν ξεχάσει. Και ήταν σημαντικό λοιπόν να ξεκινήσει ένα τέτοιο έργο που θα επιτρέψει και στην Ήπεθρο να επωφεληθεί τέτοιων έργων. Βλέπετε βέβαια το λογαριασμό εκεί πάνω. Η τοπική αυτοδιοίκηση ανέλαβε αυτό το ποσό. Από εκεί προέκυψε και η ιδέα να συμμετάσχουμε σε αυτό το πείραμα του Project Bond και εφόσον μιλάμε για πολύ υψηλή ταχύτητα τεχνολογία και μακροπρόθεσμη τεχνο... επένδυση, γιατί και το... τα ωφέλη θα αργήσουν να φανούν, Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά μπορώ να σας πω ότι προς το πάνω λειτουργεί.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 <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα γίνει σαφέστερη η εικόνα εάν εξηγήσουν οι προσκεκλημένοι μας, τους οποίους ευχαριστώ για την ενημέρωση, ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς τελικά των επενδύσεων. Για παράδειγμα, ο αυτοκινητόδρομος ανήκει στην, ομοσπονδια, στην, ομοσπονδία, στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, δηλαδή στο ομοσπονδιακό επίπεδο, στην περιφέρεια και ούτω καθεξής. Και πώς γίνεται η χρηματοδότηση του έργου. Βλέπω στη σελίδα 8 της παρουσιάσεως που βλέπω ακόμη στην οθόνη 4,38 δισεκατομμύρια κόστος κεφαλαίου του έργου. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για το σύνολο των επενδύσεων. 3,4 βλέπω προήλθαν από έκδοση ομολόγων, καλύφθηκαν δηλαδή με την έκδοση ομολόγων. Αυτά τα 562 εκατομμύρια PBCE έρχονται καπάκι από πάνω από αυτά. Δεν μου είναι απόλυτα ξεκάθαρο αυτό. Και τέλος βλέπω κάτω-κάτω, το εξηγήσατε βέβαια προηγουμένως, όταν σας ρώτησε ο κύριος Αρτουή, κάτω καθίσταται σαφές ποια ήταν η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Προϋπολογισμού. Λέει 230 εκατομμύρια. Βλέπω όμως λίγο πιο πάνω μέσα στην παρένθεση 293 εκατομμύρια που λέει ότι υποστηρίζονται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Αυτή η διαφορά από πού προκύπτει. Και το τελευταίο με ενδιαφέρει ως ε, βουλευτή μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Αν έχω καταλάβει καλά την δομή των έργων αυτών, κινητοποιούμε μέσω των ομολόγων αυτών ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία προσελκύονται δηλαδή, και υποτίθεται ότι με τους δημόσιους πόρους και στην περίπτωση αυτή ευρωπαϊκούς πόρους αναλαμβάνεται η πρώτη εγγύηση. Δηλαδή πρώτος εγγυητής είναι το δημόσιο χρήμα και μετά προστίθεται σε αυτό για την κατασκευή δηλαδή το ιδιωτικό. Εδώ δεν με ενοχλεί αυτό. Αν όμως Εφόσον όμως προκύπτουν έσοδα που καταλήγουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που φτάνουν, δηλαδή τα έσοδα από τα έργα αυτά, που τα βρίσκω στον κοινοτικό προϋπολογισμό, για να πω, δηλαδή με ειλικρίνεια, ο ενθουσιασμός μου για αυτά τα project bonds από τότε που προτριετίας στην αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού μάλωσα με το Συμβούλιο ο ενθουσιασμό μου λοιπόν έχει περιοριστεί σημαντικά. Χαίρομαι που έχουμε αυτό τον μοχλό και μπορούμε επομένω να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά εφόσον αποκομίζουμε και κέρδος, δεν έχω καμία απολύτως ιδέα που καταλήγουν στον κοινοτικό προπολογισμό. Ίσως με, με τον επόμενο πια διορθωτικό προϋπολογισμό, όπως και τα 5 δισεκατομμύρια που αναφέραμε προηγουμένως, καταλήγουν στις χώρες μέλη. Δηλαδή, εγώ ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναλαμβάνω ευθύνη με τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, δηλαδή δίνω εγγύηση, εφόσον όμως υπάρχουν έσοδα από τις επενδύσεις αυτές, τελικώς ικανοποιούνται οι Εθνικοί Υπουργοί των Οικονομικών. Πάει σε αυτούς δηλαδή το χρήμα των εσόδων ως Ευρωπαίος πολιτικός μπορώ να πάω τότε να πω στην πατρίδα μου, α κοιτάξτε ναι, συνέβαλε η Ένωση στη χρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου ε, Α7. Όμως εάν τελικώς υπάρχουν κάποια έσοδα, στην ουσία δεν λύνεται κανένα πρόβλημά μου από όσα συζητήσαμε σήμερα το απόγευμα. Ούτε για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κέρδη αυτά για την αποπληρωμή των εκκρεμών χρεών μας, ούτε καθεξής. Δηλαδή το μόνο, ο μόνος που χαίρεται τελικά είναι ο υπουργό Οικονομικών. Ε, εντάξει, είναι ένα ευγενές, ένας ευγενής πολιτικός στόχος, αλλά τι να πω, εμένα δεν με χαροποιεί ιδιαίτερα και το λέω ειρωνικά. Δηλαδή, εάν προκύπτουν κάποια έσοδα από τις επενδύσεις αυτές, θα ήθελα να φτάσουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και όχι για τους λίγους μήνες μέχρι το τέλος του έτους όπου θα επιστραφούν στις ε, χώρες μέλη. Γνωρίζω ότι υπάρχουν για παράδειγμα στα ανακυκλούμενα ταμεία ορισμένα χρήματα τα ε, οποία έγινε μια φορά μονάχα αυτό καμιά φορά είναι και πολύ δύσκολο να γίνει κατανοητή, κατανοητός μάλλον αυτός ο χρηματοπιστωτικός μηχανισμός που εφαρμόζουν και τα Εθνικά Υπουργεία Οικονομικών. Αν μπορείτε να ρίξετε κάποιο φως θα σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Επιτρέψτε μου τώρα να υποβάλω κάποια ερωτήματα. σε πρόκειται στον κ. Γκάιερ. Πρόκειται για επενδύσεις ιδιωτικού ή δημοσίου. Οι δε δαπάνε, οι πόροι που έχουν δεσμευτεί και χρηματοδοτούνται από αυτό είναι δεν είναι δαπάνε δημόσιε και αν δεν είναι δημόσιες δαπάνε, σε αυτή την περίπτωση δεν αναδύεται μία υποψία Ε, του ότι αυτό χρησιμοποιείται σαν παραθυράκι για να ξεφύγει από τη ρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας. Αλλιώς, ποιος είναι ο κίνδυνος για τον δανειστή. Επίσης, τελικά, τι ωφελεί η εγγύηση των 230 εκατομμυρίων από τον κοινοτικό προπολογισμό, γιατί από ό,τι κατάλαβα, οι σχεδίες πράξεις δεν έχουν γίνει ακόμα. Θα γίνουν αργότερα φέτος και το 2016. Αυτά 230 εκατομμύρια κατεβλήθησαν από τον κοινωτικό προπολογισμό ή όχι. Η κυρία Καλβενίου μπορεί να μα πει ότι μας πει αν αυτά ε, ήταν μια πληρωμή του προπολισμού ή όχι. Και από ποιο κονδύλιο. και αυτό που ο κύριος Κόλμελ. Ποια είναι η προσθέμενη αξία αυτών των ομολόγων έργων. Το κάνουμε για να λέμε ότι κάτι κάνει η Ευρώπη, κάτι κάνει η Τράπεζα Επενδύσεων. Όφελούν τελικά. Εάν οι οφειλέτες είναι τοπικές περιφερειακές αρχές που έτσι αναλαμβάνουν να κατασκευάσουν αυτοκινητόδρομο ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τελικά αυτά τα 230 εκατομμύρια τι ρόλο παίζουν. Αν θέλετε απαντήστε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριο Μπούρκαρτ Σμιτ. Πλήθος θεμάτων όπου μπορούμε να τοποθετηθούμε λοιπόν και εμείς. Πρώτα για την διαφάνεια για την πρωτοβουλία των ομολόγων έργου. Στο τμήμα το δικό μου της παρουσιάσεως επεσήμανα ότι αφενός υπάρχει η αξιολόγηση που είναι πρόσβασιμη και στο κοινό της πρωτοβουλίας αλλά και από τότε που τέθηκε σε ισχύ ο νέος δημοσιονομικός κανονισμός Υποβάλλει έκθεση. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δύο σκέλη της αρχής του προϋπολογισμού έκθεση για την χρήση των χρηματοδοτικών μηχανισμών. Και ο ένας από αυτούς τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, ένας από αυτούς είναι βεβαίως και η πρωτοβουλία. Δεύτερο, τονίζω ότι τα 230 εκατομμύρια που είδατε στην διαφάνεια προέρχονται από τρεις διαφορετικές, από τρεις διαφορετικά κονδύλια του προϋπολισμού από την τελευταία χρηματοδοτική προοπτική, όπου έχει συμφωνήσει ο νομοθέτης και από αυτά τα κονδύλια του προϋπολογισμού λαμβάνονται τα χρήματα τα οποία διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε ένα λογαριασμό, Τρόιχαντ, που κατατίθεται εκεί για να διασφαλίζει τη χορήγηση εγγύησης. Με ταυτόχρονη εξασφάλιση ότι ο προϋπολογισμός δεν ευθύνεται για παραπάνω από τα 230 εκατομμύρια στα οποία έχετε συμφωνήσει εσείς. Μετά τέθηκε το ερώτημα τι συμβαίνει εάν διακόπτει ο πρόεδρος. Τα 230 εκατομμύρια λοιπόν δόθηκαν σήμερα. Άρα η ΕΤΕ έχει στη διάθεσή της τα 230 εκατομμύρια. Όχι, δεν έχουν καταβληθεί. Δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το ποσό. Καταβάλλεται αναλόγως με την πορεία των έργων. Δηλαδή ποια έργα υπογράφονται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι ερώτηση του Πρόεδρου χωρίς μικρόφωνο. Επαναλαμβάνει. Ε, τα έργα αυτά θα προχωρήσουν 2015 και 2016, άρα δεν έχει γίνει ακόμα μεταφορά του ποσού αυτού. Ο έτερος των προσκεκλημένων, αν μου επιτρέπετε. Ορισμένα, μάλλον τα έργα για τα οποία σας μίλησα, όλα έχουν αρχίσει. Ορισμένα είναι λειτουργικά, ορισμένα είναι υποκατασκευή. Όλα τα παραδείγματα που σας ανέφερα σήμερα λαμβάνουν χώρα τα έργα αυτά σήμερα. Αυτή η εγγυητική επιστολή έχει εκδοθεί για όλα τα έργα. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αναλάβει κίνδυνο για όλα αυτά τα έργα. Και από σήμερα ή από αύριο μπορεί να καταπέσει η εγγύηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να επανέλθουμε για να σας εξηγήσουμε και την τελευταία τεχνική λεπτομέρεια για το πώς γίνεται η δέσμευση των 230 εκατομμυρίων, πώς περνάει δηλαδή σε μια χρηματοδοτική ροή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω από τα 230 στα 215 έχουν περάσει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε και άλλα δύο χρόνια για να περάσουμε και άλλα έργα στο χαρτοφυλάκιο. Είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι τα ενωσιακά χρήματα αποτελούν ε, τον πρώτο θεμέλιο λίθο σε ένα χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Κάθε, κάθε φορά που μπαίνει μια νέα ε, συναλλαγή στο χαρτοφυλάκιο αλλάζει το προφίλ του κινδύνου και αυτό επηρεάζει το ποσό χρημάτων που πρέπει να φύγει από τα 230 εκατομμύρια που είναι η υποχρέωση, η ανάληψη υποχρέωσης, και να πάει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και το ποσό, διορθώνω, είναι 150 εκατομμύρια. Ο κύριος Μπούρκαρ ένα τελευταίο τώρα, τέθηκε το ερώτημα από την πλευρά σας που καταλήγουν τα χρήματα τα οποία επιστρέφουν εφόσον υπήρξαν τα έργα επιτυχή και δεν χρησιμοποιήθηκε η εγγύηση. Τα χρήματα αυτά μετά από την περάτωση της εγγυητικής φάσης διαβάζονται εκ νέου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταλήγουν στην πλευρά εσόδων του προϋπολογισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή ειδικό κονδύλιο του προϋπολογισμού στο οποίο να εμβάζονται τα χρήματα αυτά στην περίπτωση της ε, πρωτοβουλίας ε, ομολόγων έργου. Ο έντρος κύριος Απλήνεται. Να σας προσπαθήσω να απαντήσω τις ε, υπόλοιπες ερωτήσεις. Γιατί νομίζω ότι θα μπορούσαμε να τι χωρίσουμε σε τέσσερις κατηγορίες. Οπότε, αν δεν έχετε αντίρρηση, έτσι να απαντήσω. Πρώτα πρώτα τις ερωτήσεις όσον αφορά την φύση αυτού του μέσου και πώς λειτουργεί. Δεύτερον, είχαμε κάποιες ερωτήσεις ε, του γιατί να έχουμε ιδιωτική χρηματοδότηση σε έναν τομέα που η απόδοση είναι χαμηλή και επίση για την επανεχρηματοδότηση και τέταρτον ε, για το έργο Κάστορ. Οπότε Α ομοδοποιήσω έτσι τις ερωτήσεις για να σας απαντήσω. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά αυτό το ίδιο το εργαλείο, το μέσον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό το εργαλείο, το ομόλογο έργο, έχει εφευρεθεί για έναν ιδιαίτερο τύπο χρηματοδότησης που στην αργό των τραπεζών ονομάζεται χρηματοδότηση έργων ή έργο. Πολλές φορές όταν λέμε εταιρική σχέση ε, ε, δημοσίου ιδιωτικού τομέα χρησιμοποιείται σαν ε, ισοδύναμο, σαν συνώνυμο αυτό που σας είπα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν αυτού του είδους τη χρηματοδότηση για τις υποδομές όπου το δημόσιο κλείνει μια συμφωνία με κάποια ιδιωτική εταιρεία ή έναν όμιλο εταιρεών ή σύμπρεση εταιρείων τέλος πάντων κατόπιν κάποιου εξωτερικού διαγωνισμού. Οπότε, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία αναλαμβάνει η εταιρεία αυτή η ιδιωτική να χτίσει, ε, να κατασκευάσει ένα εργοϊποδομή για κάποια, κάποια περίοδο. Τώρα, αυτό λειτουργεί διαφορετικά σε κάθε χώρα ή σε κάθε κλάδο. Όμως, καταρχήν και γενικώ αυτό ισχύει. Αυτό είναι η ουσία της έννοιας την οποία τώρα συζητάμε. Και έχουμε τώρα τη χρηματοδότηση που γίνεται και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και μία από τις αρμοδιότητες και ευθύνε του ιδιωτικού τομέα είναι το να εξεύρουν τα χρήματα που χρειάζονται για να, βρουν, να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τέλο πάντων αυτό το έργο σε όλη τη διάρκεια ζωής του. Και έτσι και γίνεται. Και αυτή η χρηματοδότηση κατόπιν επιστρέφεται σε αυτούς που έχουν επενδύσει για αυτό το δικό του κεφάλαιο μέσω των ταμιακών ροών που προέρχονται από το έργο. Πολλές φορές αυτό γίνεται από τους χρήστες που ας πούμε μπορεί να έχουμε κάποια διόδια ή το σπουδαίο αυτοκινητόδρομο διόδια ε, ή μπορεί αυτού του είδου ταμικές ροές να προέρχονται από κάποιες οπληρωμές που τις κάνει το ίδιο το δημόσιο και που έχουν σχέση με το στοιχείο αυτό το περιουσιακό το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με κάποιο είδους πρότυπα. Α, σας πω ένα παράδειγμα από την ε, Βρετανία που χρησιμοποιεί πολύ αυτό το μέσο. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ σε σχολεία και νοσοκομεία. Η πρωτοβουλία αυτή για το ομόλογο διακόπτει ο πρόεδρος. Ο κύριος Κόλμερ θέλει να σας διακόψει και να σας ρωτήσει κάτι πάνω σε αυτό το σημείο. Έχετε πρόβλημα. Καθόλου, καθόλου. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να θέσω μια ενδιάμεση ερώτηση. Αν μου επιτρέπετε, απλή μου λογική μου επιβάλλει να σας κάνω μια ερώτηση κατανόησης. Μιλούμε εδώ, για παράδειγμα, για την χρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου Α7 στη Γερμανία. Αν κατανόησα καλά από αυτά που λέτε, αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι η χρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου κατέστη δυνατή διότι υπάρχουν τα ομόλογα έργου. Διότι αλλιώ η Ομοσπονδιακή Γερμανία δεν θα ήταν σε θέση να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου. Δεν κατανοώ, εξακολουθώ να μην κατανοώ πού βρίσκεται το πλεονέκτημα αυτού του μοντέλου χρηματοδότησης. Εξηγήστε μου, πού ακριβώς βρίσκεται το πλονέκτημα και υπέρ τίνος λειτουργεί. Μήπως είναι ένα κόλπο για να ανακουφιστεί το χρέος. Γιατί δίνονται αυτά τα χρήματα και αυτό το ποσό μεταφέρεται εκεί που έχει καταγραφεί, έχει γραφεί το το χρέος πώς Δεν είμαι ειδικό σε αυτού του είδους, τον στον ισολογισμό και εξυγίανση αυτών των ε, χρημάτων, αυτών των τέλος μεγεθών που είπατε. Αλλά η κάθε χώρα ασκεί διαφορετική πολιτική. Όμως το βασικό πλεονέκτημα αυτού του μέσου είναι ότι χρησιμοποιώντας αυτού του είδους το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία το δημόσιο μεταφέρει στον ιδιωτικό τομέα κάποιους κινδύνους που αλλιώς θα έπρεπε να φέρει το ίδιο το δημόσιο αυτούς τους κινδύνους. Ένα παράδειγμα είναι το ότι μέσω αυτού του εργαλείου, μέσω αυτών των νομολόγων, πάντοτε μπορεί το δημόσιο να μεταφέρει στον εταίρο του ιδιωτικού τομέα τους κινδύνους της καθυστέρησης του έργου υποδομής ή της υπέρβασης του προπολογισμού σε σχέση με το κόστος στο αρχικό της επένδυσης. Επίσης και τους κινδύνους που εμπεριέχονται στο να υπάρχει κάποιο είδου τεχνικό κουσούρι, ελάττωμα, ας πούμε ένα νοσοκομείο που τελικά δεν, έχει, δεν, δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε, δεν έχει σωστή θέρμανση, ένας ε, ε, δρόμος, ας πούμε, σε αυγεντόρμος που υφίσταται κάποια κάτω και δεν παραδίδεται οπότε θα έπρεπε. Όλα αυτά θα ήταν εκείνη που θα τους έφερε κατά την παραδοσιακή μέθοδο το δημόσιο. Όμως τώρα πασάρει αυτού του είδους τους κινδύνους κατά κάποιο τρόπο στον εταίρο του ιδιωτικού τομέα μέσω αυτού του είδους ε, της, της σύμπραξης χρηματοδότησης. Και οπότε ε, έχουμε χιλιάδες σελίδες εκθέσεων των ελεγκτικών αρχών που εξετάζουν το πώς γίνεται ε, αυτού του είδους η σύμπραξη και πώς αυτό ωφελεί το δημόσιο ε, και επίσης αντίθετα όταν διαπιστώνεται ότι δεν ωφελεί το δημόσιο με τέτοια σύμπραξη και οι κρατικές αρχές όπως ας πούμε και στην Γερμανία φυσικά και έχουν την επιλογή για το πώς θα χρηματοδοτήσουν τους αυτοκινητοδρόμους και τα άλλα έργα υποδομής και το κάνουν αυτό με σύμπραξη δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Έτσι γίνεται και αυτό να πιστεύουν ότι πιάνουν τόπο τα χρήματα. Και αυτό γίνεται επειδή μπορούν να μετακυλήσουν το ρίσκο στον ιδιωτικό τομέα. Και τώρα ερχόμαστε στο γιατί να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα του ιδιωτικού τομέα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μικρής απόδοσης. Ερχόμαστε τώρα παρακάτω στο, σε κάτι το οποίο στην παρουσίασή μου δεν το ετώνησα. Δηλαδή, όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δίνει αυτή την εγγυητική επιστολή και ενισχύει το έργο με αυτά το ομόλογα έργο, η ΕΤΕ χρεώνει για την χρήση των ομολόγων. Δηλαδή, δεν παίρνει τζάμπα την εγγυητική επιστολή η ιδιωτική εταιρεία. Πληρώνει την λογική δίκαιη τιμή. Οπότε σε κάθε περίπτωση που ο ιδιώτης εταίρος ωφελείται από τον κοινωτικό προϋπολογισμό ή άλλες φορές δεν ωφελείται. Αυτό ε, γίνεται με την εγγυητική επιστολή αλλά δεν κάνει καμία διαφορά για το, το ότι βρίσκεται πίσω από αυτό το ε, ε από αυτή την κίνηση ο κινητικός προϋπολογισμός. Γιατί αυτή εξ αρχή πρέπει να καταβάλει το τίμημα στην Τράπεζα Επενδύσεων. Και το αποτέλεσμα τη εγγυητική επιστολή είναι το ότι η έκδοση των ομολόγων έργου έχει, έχουν, έχει καλύτερη αξιολόγηση. Και το ίδιο ισχύει μετά, δηλαδή έχει καλύτερη αξιολόγηση το χρέο. Το δημιουργήσουμε για αυτό το έργο που το είπαμε γκάμπαρντ ε, το χρησιμοποιήσαμε σαν παράδειγμα και να σα πω τότε που έκλεισε αυτό το έργο είχαμε 125 σημεία βάσης από το επίπεδο αναφοράς. Αυτό ήταν η αξιολόγηση. Κάτι το οποίο ε, θεωρήθηκε πάρα πολύ αυστηρό για τέτοιο έργο. Και αμέσως μετά ήρθε ο χορηγός στην ΕΤΕ ε, και το, το δημόσιο και είπε ότι ε, πιάσανε πολύ τόπο τα χρήματά μας, ας κάνουμε κι άλλο έργο. Οπότε και μετά πήγαμε στο άλλο έργο, στο Quindemore, που έκλεισε τώρα σήμερα που χρησιμοποίησε και εκεί τα ομόλογα έργο για να βοηθηθεί. Και σε αυτό το δεύτερο έργο είχαμε ακόμα πιο αυστηρή τιμή. Πήγαμε στα, στους 110 πόντους βάσης πάνω από το, την τιμή, το επίπεδο αναφοράς. Οπότε είδαμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρηματοδότης, ο, ο ιδιώτης ε, έπρεπε να ζυγίσει τα πράγματα και αν τον συμφέρει να πληρώσει για την ηγετική επιστολή το πόσο αποζητείται. Άρα όταν έχουμε ένα έργο το οποίο ε, κερδίζει, ωφελείται από την υποστήριξη του κοινωτικού προπολογισμού, τότε ε, η τιμή της κοινωτικής αποστολής ή της ηγετικής επιστολής το τίμημα αυτό το φρόντο το φέρει και ο ιδιώτης, το φέρει και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε οι τραπέζες φυσικά λένε θα μπορούσαμε εμείς να χρηματοδοτήσουμε. Φυσικά και θα χρηματοδοτούσαν. Χαζί είναι. Ε, και φυσικά και γι' αυτό και δίνουν μάχη και ανταγωνίζονται. Ε, γιατί θέλουν και αυτοί να πιάσουν από τα χρήματά τους. Όμω, όμως ο ιδιώτης τον συμφέρει να, αντί να πάει στην τράπεζα να καταφύγει στο δικό μας εργαλείο, δηλαδή τα ομόλογα έργο. Και αντίστοιχα και το δημόσιο προτιμάει όποια λύση είναι λιγότερο δαπανηρή. Τώρα πάμε στην τρίτη ομάδα ερωτήσεων, δηλαδή για την επαναχρηματοδότηση. Μάλιστα, βεβαίω και προσπαθούμε να στοχεύσουμε ό,τι μπορούμε με αυτή την πρωτοβουλία. Τα έργα Greenfield και σας είπα κάποια παραδείγματα τέτοιων έργων Greenfield. Όμως επίσης έχουμε και Brown field έργα και αυτά χρηματοδοτούνται έτσι και είναι πολύ σημαντικός στόχος για την πρωτοβουλία των ομολόγων έργων. Δηλαδή να δούμε πόσοι κεφαλαίοι κεφαλαιαγορές θα ε, συνηθίζουν πάλι το να κάνουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις σε τέτοια έργα. Και γι' αυτό και θεωρούμε ότι η πρωτοβουλία είχε τέτοιες επιπτώσεις. Πολύ παραπέρα από τις αλλαγές που είπαμε και είδατε τις στατιστικές στην παρουσίασή μας στην αρχή. Οπότε από αυτή την οπτική γωνία ήταν χρήσιμο το ότι στην αρχή της διαδρομής υποστηρίξαμε τέτοια brownfield ε, projects, brownfield έργα. Πάμε τώρα στο έργο Κάστορ. Γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση, πάρα πολύ τεκμηριωμένη. Δηλαδή κατά πόσον εμείς επενδύσαμε στο έργο Κάστορ. 300 εκατομμύρια επενδύσαμε. Και συνολικά η έκδοση ομολόγου ήταν 1,4 δις. Εμείς 300 δώσαμε. Ο λόγος προς τούτο ήταν ότι αυτό ήταν στην αρχή της διαδρομής του εργαλείου αυτού, των ομολογών έργου και είπαμε 1,4 δις ήταν έκδοση του πάρα πολλών ομολογών και εμείς ήμασταν ένας από τους ε, λίγους ε, σπόνσορες που παίζαμε το ρόλο της άγκυρας του επενδυτή για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Ε, γι' αυτό και κάναμε την επένδυση. Και όντως ισχύει ότι το έργο Κάστορ ε, ανεκτήθη από το δημόσιο. Και γιατί αυτό. Διότι μία σειρά γεγονότων σεισμικών, γεωλογικών συνέβησαν τα οποία είχαν επισημανθεί πριν αρχίσει το έργο. Και θεωρούσαμε ότι υπάρχει πιθανότητα για ένα τέτοιος σκίνδενος ε, να, να, να Τελικά ήταν πολύ πιο έντονο από ό,τι είχε υπολογιστεί, αλλά είπαμε ότι αυτά τα, είχαν, τα είχαμε επισημάνει, να την η διαφάνεια και από την άλλη μεριά βέβαια έγινε η έκδοση των ομολόγων έργου, οπότε και θα πρέπει οποιοδήποτε επενδυτή να ξέρει όλα τα δεδομένα για να αποφασίσει αν θα αγοράσει, αν θα συμμετάσχει. Ε, όλα αυτά στο προσπέκτο, στο διεθνιστικό, δηλαδή για την έκδοση ομολόγων, τα είχαμε πει. Γίνανε αυτοί οι σεισμοί. Η Ισπανική κυβέρνηση αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση του έργου, να ανακτήσει το έργο, ε, το οποίο φυσικά και το δικαιού το πλήρω. Οπότε, ε, ποιο ήταν το δίδεγμα που αντιλήσαμε ότι όταν έχουμε χρηματοδότηση κάποιου κινδύνου, όπως και το ίδιο το πλάνο Juncker, ε, τότε οι κίνδυνοι πολλές φορές επέρχονται. Ακριβώς και αυτό έγινε και με το Κάστορ. Βεβαίως αυτό ήταν κάτι παντελώς άσχετο από τη χρηματοδότηση. Επρόκειτο για κάτι τεχνικό, κάτι γεωλογικό, για έναν κίνδυνο που είχε επισημανθεί, αλλά έγινε πολύ χειρότερα από ό,τι λέγανε οι εξπέρ. Ε, όμως ε, υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι, έτσι γίνεται με τη χρηματοδότηση των έργων. Δεν είναι δυνατόν στο, ε, στο, στο, στο πακέτο αυτό να θεωρούμε ότι δεν θα επέλθουν κίνδυνοι. Ε, έρχονται κίνδυνοι και έρχονται και ζημιές. Αναλύονται, ε, προσδοκούμε, ελπίζουμε ότι δεν θα επέλθουν οι κίνδυνοι, αλλά γίνεται. Ε, αυτό πάνε να πει χρηματοδότηση κίνδυνου. Ελπίζω απάντησα. Merci. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν ερωτήσεις. Παρακαλώ. Κύριος Μαραγκάλη. Ο κύριος Μαραγκάλη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρέπει να προσθέσω μια παρατήρηση πάρα πολύ σύντομη. Μας λέτε για γεγονότα, events. Αυτά δεν είναι γεγονότα είναι αποτελέσματα των όσων έγιναν. Πρόκειται για σφάλμα της ανάλυσης κινδύνου. Σοβερό λάθος που είχε συνέπειες οικονομικές, τεχνολογικές, περιβαλλοντικές. Ε, πρόκειται για κίνδυνο που διέτρεχαν οι πολίτες. Ε, πρόκειται για μεγάλο σφάλμα της ΕΤΕ που δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Της μετακυλεί στο δημόσιο. Η οποία βέβαια ανέκτησε ε, το έργο, της έκλεισε το έργο και το έργο κατέστη άχρηστο. Ας τα πούμε ξεκάθαρα. Λέμε για το τι έγινε στο συγκεκριμένο έργο. Είδατε τι συζητήσαμε την ε, προηγούμενη εβδομάδα. Παρουσιάστηκε το Κάστορ σαν ένα έργο το οποίο κατά των πραγμάτων ακολούθησε και προέκυψε από την έκδοση των ομολόγων έργων. Όχι, ήταν ήταν ένα ναυάγιο, μια αποτυχία, γιατί δεν μπόρεσε να κάνει αυτό που έπρεπε να κάνει η ΕΤΕ, ούτως ώστε να, προχωρήσουν, να προχωρήσει το, το, το έργο και η επένδυση. Ο κ. Κέρμελ, συντομότατη ερώτηση για το έργο Κάστορ. Εδώ στην σύνοψη που έχετε υποβάλει βλέπω μια στιγμή 200 εκατομμύρια ευρώ. Τι κρίθηκε να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το έργο αυτό ή τι θα κριθεί να πληρώσει. Δεν υπήρξε επίκληση στην εγκυτική επιστολή σε αυτό το έργο. Κανείς δεν τη ζήτησε. Bien, on va en rester là. Κατέπεσε λοιπόν η ηγετική επιστολή. Ωραία, θα μείνουμε εδώ, λέει ο Πρόεδρο. Μπορείτε ίσω να μα ενημερώσετε περαιτέρω για το επιτόκιο που εφαρμόζεται και που αποδίδεται ε, σε αυτά τα ομόλογα έργου τα οποία συνδέονται και με τους 110-115 μονάδες βάσης για να δούμε τι αυτό αντικατοπτρίζει σε ό,τι αφορά την αγορά. Γιατί κατανοώ ότι οι δικαιούχοι είναι οι δημόσιοι επενδυτές. Και παρά τη σαφήνεια των απαντήσεών σας, έχω μια υποψία ότι θα δημιουργηθούν προβλήματα στους δημόσιους ισολογισμούς. Δηλαδή, για να μην επιβαρύνουμε περαιτέρω με τέτοιες επενδύσεις τον δημόσιο κορβανά, περνάμε σε τέτοια project bonds και έτσι το γλιτώνουμε αυτό. Ποια είναι η εκτίμησή σας ε, ως προς αυτό. Μετά, καλό θα ήταν πραγματικά να δείξετε την προσθέμενη αξία των ομολόγων έργου σε σχέση με άλλους τρόπους χρηματοδότησης. Αρχίσατε με, μια, με ένα τέτοιο εγχείρημα, αλλά βλέπετε κι εσείς ότι υπάρχει ακόμα ένας σκεπτικισμός. Και θα πρέπει πραγματικά να μας το αποδείξετε για να άρετε τυχόν αμφιβολίες. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και τις εξηγήσεις σας. Είναι μια πολύ ζωντανή συζήτηση ε, για τις ε, στρατηγικές επενδύσεις. που είναι, αν θέλετε, και το τελικό αποτέλεσμα του πειράματος ε, αυτού για τα ομόλογα έργου. Θα περάσω στο επόμενο σημείο, γιατί δεν είναι εδώ ο συνάδελφος. Επομένως, θα το εξετάσουμε. Η ανταλλαγή απόψε δηλαδή, θα γίνει στις 26 Μαΐου. 28 Μαΐου ημερομηνία κατάστασης τροπολογιών και αρχές Ιουνίου η ψήφιση σε ό,τι αφορά το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Για το τμήμα της ε, τεχνικής ε, συνδρομής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, μια τέτοια συνδρομή μπορεί να μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα το μηχανισμό εκτέλεσης. Monsieur doit nous faire connaître... Ο κύριος Ταράν θα μας ε, ενημερώσει για την ε, αλληλευτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γουινέας Μπισάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, πολύ γρήγορα και σύντομα. Είναι μια καλά σορπημένη συμφωνία. 10 Λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ κατά έτος είναι οι δαπάνες. Εμείς κερδίζουμε σε αλλιεύματα, εκείνοι κερδίζουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και χρήματα. Το μοναδικό συναρπαστικό εδώ είναι ότι η συμφωνία ολοκληρώθηκε και συνήφθη μάλλον το 2012 για τρία χρόνια. Ουσιαστικά δηλαδή κάνουμε κάτι για μια συμφωνία που θα λήξει εντός λίγων ημερών. Αυτό περιγράφει πόσο καθυστερούν οι ευρωπαϊκές διαδικασίες. Κατά τη γνώμη μου, το Κοινοβούλιο θα πρέπει ε, να υιοθετεί, να εγκρίνει, να γνωμοδοτεί τέτοιου είδους ε, συμφωνίες πριν αρχίσουν να ισχύουν. Πόσο μάλλον όταν φτάνουν κοντά στη λήξη τους. Ωστόσο, στηρίζω την ε, γνωμοδότηση και με ενημέρωσαν ότι θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε τροπολογίες στην ε, καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή της Αλίας, γιατί θα υπάρξει και ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που θα συνοδεύει τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις. Όχι από ό,τι βλέπω. Τροπολογίες πριν τις 11 Μαΐου θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 22-23 Ιουνίου και καταρχήν η ψηφοφορία στην Επιτροπή Αλίας θα γίνει 15-16 Ιουλίου. Πολλά μέλη της Επιτροπής μας ε, συμμετείχαμε στην, στην αποστολή στην Ουκρανία 18, 19 και 20 Μαρτίου. και το μέλος ε, της Επιτροπής μας Αντρέας Πλένκοβιτς που είναι και πρόεδρος της ομάδας φιλίας μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωσέ Μανώλη Φερνάντες, Κλέρ Μούντι, Ινιέζε Βάιντερα, Μόνικα Βανά και Ντανιέλ Βιώτη. Κατόπιν ε, αυτής της επίσκεψης πρέπει να κάνουμε μια σύνοψη που έχει διαβιβαστεί σε όλους σας. Βρήκαμε μια χώρα που περνάει δύσκολες μέρες γιατί ασκούν σημαντικές πιέσεις στα ανατολικά της σύνορα από ρωσόφωνους πληθυσμούς ε, που καταφανώς και ε, τη χάνουν στήριξη ε, της Ρωσίας πέραν της Κρυμαίας που είναι μια μόνιμη κατάσταση και δεν τηρείται το πρωτόκολλο του Μίνσκ. Πολλοί συμμετείχαμε. Είμαστε, συγγνώμη, ε, πολλοί ήταν οι εκτοπισμένοι, πάνω από ένα εκατομμύριο 200.000 άτομα, τα οποία θα πρέπει κάποιο να τα αποδεχθεί, ε, να φροντίσει για την περίθαλψη, την παιδεία και ούτω καθεξής. Εξαιρετικά δύσκολες συνθήκε. Μια χώρα που αντιμετωπίζει και τεράστια οικονομικά προβλήματα και πρέπει να πάρει εξαιρετικά επώδυνα μέτρα και αποφάσεις για τον ε, ντόπιο πληθυσμό. Γιατί η ε, η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν κατάφερε να καταπολεμήσει τη διαφθορά και μεταξύ των πολύ σημαντικών τομέων όπου υπάρχει διαφθορά υπάρχει, υπάρχουν και τα τελωνία, υπάρχει και το ζήτημα ε, με το φυσικό αέριο γιατί τα ολιγοπόλια αυτά ε, εποφελούνται ε, της κατάστασης με το φυσικό αέριο και της διανομής του. Για να πάρει κάποιος αυτή την επιδότηση που θα μπορούσε να δοθεί σε έναν νοικοκυριό, ε, μεταφέρει κάποιος ε, την κατανάλωση της επιχείρησής του σε οικιακή κατανάλωση και έτσι γίνεται η διαφθορά. Στις μεταρρυθμίσεις που εξετάζουμε εμείς είναι η επανεξιολόγηση του κόστου του φυσικού αερίου που είναι τεράστιο εγχείρημα βεβαίω. και δύσκολα θα γίνει αποδεκτό. Υπάρχει σημαντική κινητοποίηση και η Ευρώπη συμμετέχει ενεργά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται εκεί μαζί με ικανότατες και εξαιρετικά ομάδες Επίσης είδαμε και τους ε, χορηγούς που είναι πολλοί. Σε ό,τι αφορά τον ε, συντονισμό, υπάρχει ακόμα θεματικό περιθώριο βελτίωσης, από ό,τι φαίνεται. Ορισμένοι εκπλήσονται που η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ηγείται αυτού του έργου του συντονισμού. Κανονικά πρέπει να είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης, αλλά η κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να διασφαλίσει αυτό το συντονισμό. Επίσης, ε, παρατήρησα ότι οι ομάδες μας εκεί δυσκολεύονταν να πάρουν από τις Βρυξέλλες ε, τις αναμενόμενες ε, αποφάσεις. Και αυτό δημιουργούσε προβλήματα στο εσωτερικό των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα πολλά θα μπορούσε να πει κάποιο ακόμα, όπως και να έχει το κύριο αναφέρεται σε αυτό το έγγραφο. Μπορείτε να πάρετε το λόγο για το περιεχόμενό του. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Ε, bien, si personne ne souhaite prendre la parole. Εάν δεν υπάρχει κάτι. Si Επιτρέψτε μου να επιμείνω στο εξή. Αν θεωρείτε ότι έχει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ηγηθεί αυτή τη διαδικασία ή όχι. Για να είναι απολύτω αποτελεσματική. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες τώρα. Σας ε, παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες σας ε, ε, στο μηχάνημα. Να κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο. Euh,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 σαν Nous reprenons nos travaux puisque l'heure est venue. ξεκινήσουμε λοιπόν. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στι ψηφοφορίε. Πριν ψηφίσουμε, παρακαλώ α ελέγξουμε πρώτα τα... κάρτε σα. Παρακαλώ ψηφίστε. πέρας. Χαιρετίζω όσους ε, υπερψήφισαν. <laughs> Βλέπω ότι κάποιοι καταψήφισαν και άλλοι προτίμησαν να απόσχουν. Ωραία. Όλα βαίνουν καλώ. Εσείς τι κάνετε, ψηφίζετε υπέρ ή κατά. Κάποιος δεν ψήφισε. Ναι, τον βρήκαμε τον ένοχο, ο πρόεδρος. Ωραία. Πρώτα θα ψηφίσουμε για την έκθεση που αφορά την αξιοποίηση των διατάξεων της συνθήκης Λισαβόνας. Είχα την τιμή να σας ε, υποβάλω αυτή την ε, έκθεση γιατί μου την είχατε αναθέσει. Τροπολογία 8, στον 1, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 9. Αποσύρεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική υπαριθμών 1. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 4α νέο. Τροπολογία 16. Η προφορική τροπολογία του κυρίου Τάγκ έχει ενσωματωθεί στο δεύτερο τμήμα. Το πρώτο τμήμα, notes that, μέχρι by the council. Για το πρώτο τμήμα λοιπόν. Υπέρ. Πρώτο τμήμα. Εγώ δεν είδα τίποτα ακόμα. Πρώτο τμήμα. Με την προφορική τροπολογία. Αρνητική γνώμη του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Budgetary explanation. Και που. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Στην παράγραφο 4β. Α, Επειδή υπερψηφίστηκε 15. Παράγραφος 5, τροπολογία 18, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 20 αποσύρεται, όπως και 21. Συμβαστική 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 6α νέο. Τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνώ στις ιδεολογικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Με προφορική τροπολογία.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 Ας ψηφίσουμε επί του συνόλου της νομοδότησης. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση. 29 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Και δεν υπάρχουν αποχές. Τώρα για την έκθεση του κυρίου Ντενανό. Για το σύνολο του κειμένου. Που εγκρίνει την εταιρική σχέση. Αρχικά επί της συμφωνίας. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Και για τη γνωμοδότηση του κύριου Ντενανού. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 30 ψήφοι υπέρ, 1 κατά, δύο αποχές. Μετά, έκθεση Χωσέ Μανουέλ Φερνάντες για το πράσινο ευρωτήρι. Sur, euh, sur, sur l'accord. Για την συμφωνία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται και για τη γνωμοδότηση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 ψήφοι υπέρ, μία κατά, 5 αποχές. <laughs> Sur le budget, budget 2015. του 2015. Δήμα 3. Η κυρία Γκορδία Ζαμπάλ. Και απροβαρό Θα πρέπει να εγκρίνουμε πρώτα αυτά τα 40 εκατομμύρια για την ανθρωπιστική αλλά για τον Νότιο Σουδάν και τις όμορες χώρες και υπάρχει ανθρωπιστική κρίση πάρα πολύ εκτοπισμένη οπότε και υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ε, πείνα κλπ. Μιλάμε και 40 εκατομμύρια ευρώ τόσο ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Να ελαφρύνουμε κάπως την κατάσταση. Και η άλλη μεταφορά πόρων είναι πάλι ανθρωπιστική βοήθεια, 15 εκατομμύρια ευρώ σε αυτή την περίπτωση για να βοηθήσουμε την Ανατολική Ουκρανία όπου και εκεί είχαμε ε, εσωτερικά εκτοπισμένους αλλά και αυτοί χρειάζονται τη βοήθεια του κινητικού προπολογισμού και έτσι θα βοηθήσουμε το πρόγραμμα βοήθειας στο ΟΗΕ. Βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας. Οπότε προτείνω να εγκριθούμε και τις δύο προτάσεις. Να ψηφίσουμε συνολικά για να μην υπάρξουν προβλήματα. Ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Να ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 27 ψήφι υπέρ Μία κατά, δύο εποχές. Madame Holmeyer, est-ce qu'il y a des... Κυρία Χολμάιερ, υπάρχουν μεταφορές κατόπιν αιτήματός σας? Il n'y en a pas Όχι. Alors on va passer à la politique du patrimoine. Ας περάσουμε στην πολιτική κληρονομιάς λοιπόν. Να σας δώσουμε το λόγο. Ευχαριστώ. Σήμερα καλούμεθα να ασχοληθούμε με ένα κτίριο. Θέμα που μας είχε απασχολήσει στο τέλος του προηγούμενου έτους και εμείς είχαμε εγκρίνει τότε μεταφορά 22 εκατομμύριων ευρώ για λογαριασμό της Κομισιόν, διότι το κτίριο Ζαμονέ 1 είναι μολυσμένο με αμίαντο και δεν είναι δυνατόν να εγγυηθεί κανείς ότι δεν θα υπάρξουν βλάβες υγείας του προσωπικού. Και ο κίνδυνος αυτός βεβαίως δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν προέβη σε έρευνες γιατί για να βρει τόσο γρήγορα, τόσο γρήγορα κτίριο για 1800 και κάτι συνεργάτες δεν είναι τόσο εύκολο. 200 συνεργάτες κατανεμήθηκαν σε τέσσερα προϋφιστάμενα κτίρια σε προϋπάρχοντα γραφεία που ήταν διαθέσιμα, χρησιμοποιεί επίσης τηλεεργασία κλπ. Άλλους 200 βρήκε προσωρινή λύση και παραμένουν περίπου 640 συνεργάτες. Για 6 χρόνια πρόκειται να μισθωθούν τρία κτίρια. Ο Δήμος του Λουξεμβούργου εμφανίστηκε πολύ γενναιόδωρος και προσφέρει ένα κτίριο ολόκληρο και καλείται η Κομισιόν να πληρώσει μονάχα τα λειτουργικά έξοδα. Εκεί πραγματικά αξίζει να ευχαριστήσει κανεί τον Δήμο Λουξεμβούργου, διότι μπορεί το κτίριο αυτό να στεγάσει 516 συνεργάτες. Δεύτερο κτίριο, μπορεί να καλύψει 588 ε, συνεργάτες πάλι για μια εξαίτια και άλλο ένα τρίτο πάλι για εξαίτια. Βεβαίως εφόσον γίνονται μισθώσεις για έξι χρόνια αφενός υπάρχει προβλέψιμο της μισθώσεως, από την άλλη μεριά είναι κατεσπαρμένοι οι συνεργάτες. Υπάρχει το ενδεχόμενο το κτίριο CAD να είναι έτοιμο νωρίτερα το δικό μας κτίριο. Αλλά αυτό διαθέτει μονάχα 300 θέσεις. Άρα οι υπόλοιποι 200 συνεργάτες θα πρέπει να μείνουν κάπου αλλού. Ίσως στα υπόγεια του κτίριου Ντρόσπαχ σε διάφορα μέρη. Αυτά βεβαίως είναι απαράδεκτα. Άρα δεν έχουμε άλλη λύση παρά να δεχθούμε την μίσθωση του κτιρίου Αριάν του οποίου εκμισθωτή θέλει να το μισθώσει ολόκληρο, αρνείται να το μισθώσει μόνο εν μέρη. Αυτές είναι οι επιλογές, διότι πρέπει οι συνεργάτες να μπορέσουν να εγκαταλείψουν τα άλλα κτίρια σύντομα. Αυτό ω συνέπεια έχει. Αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υπολογίσει ένα κόστος μέχρι 200 εκατομμύρια. Κάτι που μας είχε τρομάξει στην αρχή. Τώρα έχει κατέβει στα 112-113 εκατομμύρια σε αυτό ε, συνυπεύθυνο είναι βέβαια και το κράτος του Λουξεμβούργου. Προσφέρει βέβαια ένα κτίριο που βαρύνει μόνο το λειτουργικό κόστος. Τα λειτουργικά κόστη είναι συνολικά 13 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Συμπληρώστε σε αυτά το κόστος της μεταφοράς 650.000 και ετησίως διάφορα έξοδα της τάξης συνολικά του 2,15 εκατομμυρίων. Ο πρώτος Διακόπτη δεν έχει μικρόφωνο, δεν τον ακούμε. Καλά, θα προσπαθήσω να τα λέω πιο αργά, αλλά η δυσκολία είναι ότι είναι τρία τα κτίρια και όσο περισσότερο σας εξηγώ, καλά θα προσπαθήσω για χάρη των μεταφραστών να τα πω πιο αργά. Οι μεταφραστές ευχαριστούν την κυρία Χολμάρη. Το δεύτερο κτίριο τώρα, το κτίριο Αριάν, εκεί το ετήσιο μίσθωμα θα είναι της τάξεως των 4,6 εκατομμυρίων με αύξηση ανά 1,9%. Fit out, εξοπλισμός δηλαδή, 6,49 εκατομμύρια υποθέτουμε. Συνολικά δηλαδή περίπου 7 εκατομμύρια. 600 περίπου χιλιάδες εξοπλισμός ε, για ηλεκτρονικές ε, εφαρμογές, συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος 2,5 εκατομμύρια και με τη μαριθμική αναπροσαρμογή της τάξης του 1,9%. Αυτό θα φανεί βέβαια αν επαληθεύεται. Για 6 χρόνια πάλι το κόστος της Αριάν ενέρχεται σε 55,3 χωρίς να, να λέγει τι ακριβώς εννοεί. Το άλλο κτίριο, Ακολίτ, 43 εκατομμύρια, 4,3 μίσθωμα που θα πρέπει να πληρωθεί. Συμπεριλαμβάνεται πάλι το 1,9% της αριθμικής αναποσαρμογής, ώστε για τα 6 χρόνια θα φτάσει περίπου τα 25 εκατομμύρια. Εξοπλισμός, 3,3%, 10% συν πλήν, 3,6% λοιπόν ο σχεδιασμός για να μην μείνουμε πολύ έξω για τα fit out περίπου 600.000 για την μετακόμιση περίπου το ίδιο ποσό όπως ανέφερα προηγουμένως δηλαδή περίπου 250.000 όπως και για τα άλλα κτίρια ετήσια λειτουργικά κόστη περίπου 1,9 εκατομμύρια τη μαριθμική αναπροσαρμογή 1,9% ανά έτος. Θα δούμε τώρα αν θα είναι 1,9% ή 1,7%. Θα φανεί αυτό στα χρόνια όπου θα λειτουργήσει η τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος. Πιο συγκεκριμένα τώρα, για τον προϋπολογισμό. Εμείς έχουμε μεταφέρει 22 εκατομμύρια. Μας μένουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια από τα έξοδα του Ζαμονέ έχουμε ακόμα 6 εκατομμύρια. Από την μεταφορά συνολικά από τα 47 εκατομμύρια έχουμε 22 εκατομμύρια και άλλα 25 εκατομμύρια διαθέσιμα τα οποία είναι ακόμα εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό. Ένα στιγμή να βρω το σχετικό σημείωμα. Αυτό σημαίνει ότι τα 22 εκατομμύρια και τα 12 εκατομμύρια για το κόστος του 2015 τα 22 εκατομμύρια χρησιμοποιήσουμε τα 22 εκατομμύρια για να προσπαθήσουμε πάλι να μεταφέρουμε άλλα 21 εκατομμύρια για το 2016 διότι στον προϋπολογισμό λόγω του ότι διαθέτει δωρεάν ένα κτίριο το Λουξεμβούργο και επομένω το κόστος αυτό δεν βαρύνει το 2015 μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για το 2016 αυτό μειώνει κάπως την πίεση για το 2016 συνολικά το κόστος μέχρι το 2021 θα είναι 112,8 εκατομμύρια, δηλαδή 113 σχεδόν. Και η ιδιαίτερη επιβάρυνση είναι μεταξύ 2017 και 2019. Και όταν θα επανέλθουν στο κτίριο Ζαν Μονέ, τότε μειώνονται τα ετήσια έξοδα πάλι θα σας ε, κοιτάξω μια στιγμή στον πίνακα, καταλήγουμε πάλι στα 33 εκατομμύρια ανά έτος το 2022, 21-22. Αλλά η ενδιάμεση φάση όπου de facto θα πρέπει να γίνεται διπλή δουλειά και επομένως δημιουργείται έξτρα κόστος λόγω του ότι μισθώνονται και άλλα τρία κτίρια Λοιπόν, αυτή η διάμεση φάση ανέρχεται στα 113 εκατομμύρια. Πάλι καλά που δεν είναι 200, αλλά και 113 εκατομμύρια πολλά είναι. Δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς όμως, αν δεν θέλει να διακινδυνεύσει η υγεία των εργαζομένων. Στο κτίριο Goldbell συζητούμε αυτή τη στιγμή με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να μετακινηθεί στο κτίριο Goldbell νωρίτερα γιατί στο κτίριο Καντ, Κόναντ Αντενάουερ δηλαδή, οι άμεσοι γείτονες, οι, άμεσα, οι άμεσοι γειτονικοί χώροι ήταν υποχρεωτικό να εκενωθούν γιατί γίνονται εργάσεις. Τώρα βεβαίως οι εργασίες προχωρούν ταχύτερα και θα μπορέσουν να επανέλθουν οι συνεργάτες μας ταχύτερα στο κτίριο Αντενάουερ και στο γειτονικό κτίριο. Αφού τώρα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, χάρη στο ΕΦΣΙ, ψάχνει να βρει τώρα άλλο κτίριο, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε με την Τράπεζα Επενδύσεων, έτσι ώστε ενδεχομένως να εξοικονομήσουμε το κόστος αυτό και τελικά να μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό βεβαίως για τον προϋπολογισμό του Κοινοβουλίου, διότι ο προϋπολογισμός της Κομισιόν επιβαρύνεται με το ποσό των 113 εκατομμυρίων. Αυτή ήταν η προσπάθειά μου να συνοψίσω ένα πολύ περίπλοκο ντοσιέ. Χωρίς να σας ταλαιπωρώ για 15 με 20 λεπτά. ευχαριστώ να με ρωτήσετε ό,τι θέλετε. Θαυμάσια τα καταφέρατε, λέει ο πρόεδρος. Την επόμενη φορά ίσως θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδου προβολή, ούτω ώστε να μπορούμε να δούμε του πύργου, τα ακίνητα βεβαίω, να ευχαριστήσουμε και την κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου για όλα όσα έθεσε στη διάθεση του Κοινοβουλίου, ούτω ώστε να μειωθούν τα έξοδα. Ε, Κύριε Χόρμαϊ, αν θέλετε να έχετε μια επισκόπηση, κοιτάξτε στη σελίδα 14 του εγγράφου, θα δείτε ένα πίνακα που δείχνει με καθαρό τρόπο το πόσο περίπλοκες είναι οι δαπάνες τελικά. Οπότε, η εισηγήτρια ζήτησε να μάθει αν έχετε κάποια ερωτήματα ή κάποιες παρατηρήσεις. Κύριε Ντεπρέ, το 2016 είχαν εγγραφεί αυτά τα 16 εκατομμύρια. Δεν είμαι στέση να απαντήσω, πρώτα. Θα πρέπει να μου έχετε πει ότι θα με ρωτήσετε από πριν. Θα ήταν προς έκπληξη αν κάτι προβλεπόταν. Γιατί το λέω αυτό, για να <laughs> καθυστερήσει ψηφοφορία. Ε, Κύριε Χόλμα, για το 2015 δεν αναμένουν δυσάρεστες εκπλήξεις των κύριο Ντέπρε. Για το 2016, στο τέλος του έτους, θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταφορά πιστώσεως 21,6 εκατομμυρίων, ώστε για το 2016 να είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Το 2016 λοιπόν θα χρειαστούν πια, εφόσον γίνει αυτό, μόνο 4 εκατομμύρια πρόσθετα. Το 2016 λοιπόν τα πράγματα είναι σχετικά χαλαρά. Για το 2017 πια θα χρειαστεί να ξανακάνουμε άλλη προετοιμασία. Αυτά για το 2016 και 2017. Oui, pardonnez-moi, c'est pas, c'est la Commission, c'est pas, c'est pas le Parlement. με, αλλά είστε Επιτροπή, όχι το Κοινοβούλιο. Τι καλύτερο κομπλιμέντο από την απουσία ερωτήσεων, κύριε Χολμάγερ. Σημαίνει αυτό ότι η ομιλία σας ήταν άκρος διαφωτιστική. Θέλετε να ψηφίσουμε τώρα. Bon. Comme sont des transferts, il faut voter. Πρόκειται για μεταφορά πιστώσεων. Πρώτα πρέπει να ψηφίσουμε. Α, αρκεί η ανάταση χειρό, μάλιστα, λέει και η Γραμματέία. Καλά. Η ανάταση του χειρό, συγκρίνεται τα όσα πάρει ο κ. Χολμάκη, μάλιστα. Ποιοι είναι κατά. Μία ψήφος, κατά, αποχέ. Τέσσερι απόχέ. Le Επομένη έκθεση. αναβάλλεται για δύο εβδομάδες γιατί έχουμε προς την υπηρεσία Λίζα πολλά ερωτήματα. 26 Μαΐου η επόμενη συνεδρίαση. Ah oui, oui. Mais j'ai noté que vous étiez tous d'accord pour le report de deux semaines euh, <laughs> du rapport que ma... Ah, symphonie de συμφωνείτε για αυτή την ε, αναβολή του θέματος κ. Σχολμάγερ. Δύο εβδομάδες anavolie. 26 Μαΐου στις Βρυξέλλες και 27 Μαΐου στις Βρυξέλλες. 27 Μαΐου είναι έκτακτη συνεδρίαση. Παρουσίαση το σχεδίο προϋπολογισμού του 2016 της, ε, της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος πάντων. Διάφορα τίποτα πέρα συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Oui, oui, oui, oui, oui.